Well, ladies and gentlemen, it's past. Κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει πέντε λεπτά από την ε, προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασής μας, επομένως πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά. Θα συζητήσουμε το, τις επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να καθοσορίσω όλους τους ε, συμμετέχοντες σε, αυτό το, σε αυτή το workshop, σε αυτή τη συζήτηση. Μου είχαν πει ότι θα γεμίσει αυτή η αίθουσα που κλείσαμε, μία από τις μεγαλύτερες. Δεν έχει γίνει αυτό ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια συζήτηση ε, αναλυτική με τους ε, συμμετέχοντές μας από κοντά, κάτι που είναι σημαντικό. Μπορούμε να συζητήσουμε διάφορα θέματα, ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι το ενεργειακό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα συστήματα των μελών, κρατών μελών είναι διασυνδεδεμένα. Υπάρχουν συνδέσεις άμεσες ηλεκτρική, ε, ηλεκτρικής, ε, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ Γαλλίας και Ολλανδίας για παράδειγμα υπάρχουν αγωγοί και εντός της ε, υπηρετικής Ευρώπης έχουμε επίσης αγωγούς με την Νορβηγία και έχουμε επίσης και μεταφορικά ε, συστήματα. Έχουμε το τούνελ της Μάνχης επίσης. Δεν φαντάζομαι ότι θα το κλείσουμε μετά το Brexit. Παρεπιπτόντως έχει μείνει λιγότερο από ένας χρόνος μέχρι το Brexit και ο στόχος της σημερινής μας συζήτησης είναι να συζητήσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει για την ενέργεια και ε, την τιμή της ενέργειας για το υπόλοιπο 27 κράτη ε, της Ένωσης για αποχώρηση του ΕΒ. Βασιλείου. Πρακτικές πληροφορίες. Έχουμε μια μισή ώρα ε, για την συζήτηση, για αυτό το workshop και προετοιμαστείτε να είστε έτοιμοι γιατί η συνεδρίαση μεταδίδεται και μέσω του διαδικτύου έχουμε web stream. Οι παρουσιάσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής ε, Ήτρε και ε, μια περίληψη των διαμυθέντων στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο στους ομιλητές με... και θα σας ζητήσω να τηρήσετε ένα χρόνο ομιλίας 10 λεπτών. Έχω διαπιστώσει ότι οι πολιτικοί δεν τα καταφέρνουν να κρατάνε το χρόνο ομιλίας, να τον τηρούν. Αυτά τα 10 λεπτά, 5 λεπτά, ό,τι όριο και να τους βάλεις. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τεχνικά θέματα τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά. Θα δω λοιπόν ε, αν όντως είστε μηχανικοί από το πόσο καλά θα τηρήσετε το όριο χρόνου. Μετά από τους συμμετέχοντες στο πάνελ θα έχουμε και συζήτηση. Θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις από τα μέλη της Επιτροπής και από το κοινό. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω αν γίνεται ή ανάλογα ίσως δίνω το λόγο σε κάθε μιλητή για να απαντά κατευθείαν μετά την ερώτηση που του ετέθη. Θα πρότεινα λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ταλιαπέτρα, τον πρώτο μας ομιλητή, ο οποίος θα μας δώσει μια συνολική ε, εικόνα του, πιθανών, του πιθανού αντικτύπου του Brexit στο ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Τελιαπέτρα είναι ειδικό σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, είναι ειδικό επίσης σε θέματα διεθνών αγορών ενέργειας ε, και τις ενεργειακές σχέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και με, στην Ευρω... Ε, Μεσογειακή περιοχή. Είστε επίσης μέλος στην Οικονομική ε, Ένωση της Euromed και σας δίνω μέσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σίμωνα Τελιαπέτρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που θα μου δώσει την δυνατότητα να συζητήσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει το Brexit στις αγορές ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήθηκε από την Επιτροπή Ήτρε να διεξάγει μια μελέτη έτσι ώστε να αντιληφθούμε καλύτερα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. αυτό γιατί έχει γίνει μια σχετική μελέτη για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει όμως να δούμε και εμείς ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τους πολίτες και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα παραμείνουν μετά το Brexit όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας. Και για να διεξάγουμε αυτή τη μελέτη εξετάσαμε οκτώ θέματα τα οποία θα σας αναπτύξω σήμερα. Είδαμε πρώτα απ' όλα την ε, σχέση, τη μελλοντική του ε, Ηνωμένου Βασιλείου με την αγορά ε, ενέργειας της Ευρώπης, την, τη χρηματοδότηση που θα υπάρχει, την σχέση με τις ρυθμιστικές αρχές. Είδαμε επίσης πώς θα προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή χωρίς την συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Είδαμε επίσης το σχετικό και σημαντικό ζήτημα της ασφάλειας, της ενεργειακής όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Και πιο συγκεκριμένα ποιος θα είναι, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη πιο συγκεκριμένα ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για τις επιχειρήσεις στην Ιρλανδία. Να σας πω εξ αρχής ότι δεν διαπιστώνουμε να ε, προβλέπεται να υπάρξει μια σημαντική επίπτωση του Brexit στα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια. Θεωρούμε ότι ε, είτε με είτε χωρίς τον νομονοβασίλειο τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους για την κλιματική αλλαγή και να κρατήσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια. Τούτου λεχθέντος. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να επιληθούν ε, με διαπραγματεύσεις πολλά, ε, ε, πολλές λεπτομέρειες, πολλά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις που θα έχει το Brexit για το ενεργειακό σύστημα της Ιρλανδίας. Αυτό θεωρούμε από τη μελέτη μας ότι είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Θα εξετάσω λοιπόν αυτά τα οκτώ θέματα στα, οποία αναφέρθηκα ε, το ένα μετά το άλλο, ξεκινώντα πρώτα απ' όλα από την πρόσβαση που θα έχει το Ηνωμένο Βασίλειο στην ενεργειακή αγορά του, Ευρωπαϊκή της, Ω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέλος του ΠΟΕ δικαιούται να εξάγει και να εισάγει ενέργεια ε, άνευ δασμών με άλλα, ε, προς άλλα ε, μέλη θεωρούμε ότι είναι και προς αμοιβαίο όφυλος και, του ΕΒ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρεθεί ένας διακανονισμός έτσι ώστε να συνεχιστούν οι ανταλλαγές ενέργειας που ήδη λειτουργούν και υπό αυτή την έννοια δεν περιμένουμε να, υπάρξουν, ε, να υπάρξει κάποια αναστάτωση ε, εξαιτία του Brexit. Ωστόσο, από τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον δεν θα συμμετέχει στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ούτε θα είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί τους κανόνες, θα μπορούσε να επιλέξει να μην συμμετέχει πια στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα βελτιστοποίησης, το οποίο θα είχε επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης της ενέργειας. Κατά την άποψή μας αυτό θα είχε ε, σε μεγαλύτερο βαθμό δυσμενή αποτελέσματα για το Ηνωμένο Βασίλειο παρά για την Ευρώπη των 27 Κατά τα άλλα, όσον αφορά την φορολογία της ε, ενέργειας, δεν θεωρούμε ότι το Brexit θα έχει κάποια επίπτωση μιας και ε, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επενέβαινε σε αυτό. Όσον αφορά τώρα την προσφορά, την, την ε, δυνατότητα χρήσης ε, κονδυλίων, που, ποια θα είναι διαθέσιμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει μικρότερη πρόσβαση, πιο περιορισμένη πρόσβαση σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία όπω το Επιδυτικό Ταμείο, το Connecting Europe, τον Ορίζοντα 2020 και άλλα. Ωστόσο, ε, μην ξεχνούμε ότι αυτά τα ζητήματα συνεχίζουν να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση και ένα ε, σημαντικό στοιχείο είναι η σχέση που θα κρατήσει το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων. Δεν συνδέεται προφανώ μόνο με την ενέργεια, αλλά γενικότερα με τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και είναι ένα σημαντικό χαρτί, αν θέλετε, στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση σε στην, στις ρυθμιστικές αρχές. Θεωρούμε ότι δεν θα αλλάξουν ουσιαστικά οι ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου και τη λειτουργία και στις τέσσερις μεγάλες ρυθμιστικές αρχές ή συνδυασμούς ρυθμιστικών αρχών που έχουμε, Acer, CER, ENSO και ENSOC. Ε, θα αλλάξει βεβαίως η συμμετοχή εκπροσώπων, όμως εάν υπάρξει σχετική συμφωνία, θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει ίσως με κάποια άλλη ιδιότητα σε αυτούς τους σε αυτούς, οργανισμούς, σε αυτά τα όργανα, όπως εξάλλου συμβαίνει και με άλλες χώρες ε, συνδεδεμένε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο ήταν πολύ ε, σημαντικό και υψηλά στις προτεραιότητες της ε, δημόσιας συζήτησης ήταν το ερώτημα του κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους της για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την κλιματική αλλαγή. Κατά την άποψή μας, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίσει να ακολουθεί τους στόχους που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, θα μπορούσε να συζητηθεί η συμμετοχή του και στις ε, δομές ε, συντονισμού και διακυβέρνησης των στόχων αυτών. Εάν πάλι επιλέξει να μην ε, ε, τηρήσει αυτέ τι δεσμεύσει, αυτού του στόχου. Και πάλι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προσαρμόσει τι δικέ τη δεσμεύσει και του δικού του στόχου έτσι ώστε να πετύχει τον γενικό. Ε, η αλλαγή δεν θα είναι δραματική για την Ευρώπη των 27. Στον αφορά το σύστημα εμπορία δικαιωμάτων εκπομπή ρήπων γνωρίζουμε ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε βραχυπρόθεσμο ε, ε, ε, στάδιο θα δημιουργήσει ένα πλεόνασμα δικαιωμάτων εκπομπής. Όμως μακροπρόθεσμα αυτό θα σβήσει. Όσον αφορά τώρα τους κανόνες για την ενεργειακή ασφάλεια και όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και όσον αφορά το φυσικό αέριο, δεν θεωρούμε ότι όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια θα υπάρξει καμία επίπτωση για την Ευρώπη των 27 από τον Brexit. Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ μικρή. Είναι μικρότερο του 1% της συνολικής κατανάλωσης. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το φυσικό αέριο η εμπορία είναι μικρή. Όμως, και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, υπάρχει σημαντική εμπορία, ε, σημαντικό εμπόριο φυσικού αερίου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας η οποία Ιρλανδία εισάγει το 56% του φυσικού αερίου που καταναλώνει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμπέρασμα η ενεργειακή ασφάλεια όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο δεν θα επηρεαστεί για τους 27 από το Brexit, όμως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, θα πρέπει να δούμε πιο επισταμένα την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ιρλανδία. Πυρηνικά, πυρηνική ενέργεια. Εδώ βρίσκεται το ερώτημα του ποια θα είναι η μελλοντική σχέση της ε, Ευρατόμ με το, με το Βασίλειο. Γνωρίζουμε ότι ήταν ξεκάθαρο στο, στη Λευκή Βίβλο για το Brexit και ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρο μετά από τη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων και στην Βουλή των Λόρδων ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούσε ότι θέλει να αποχωρήσει και από την Ευρατόμ παρά το γεγονό ότι είναι ένα ξεχωριστό διεθνή οργανισμό με ξεχωριστή συνθήκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι. Και παρόλο που συζητήθηκε το θέμα, γιατί να μην παραμείνουν αφού είναι ένα τεχνική φύσεω οργανισμό, Επιθυμεί λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει και από την Ευρατόμ. Κατά την άποψή μα, λοιπόν, δεδομένε αυτής της απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να, ε, τεθούν, ε, να, να, βρεθεί, να ε, βρεθούν συγκεκριμένε πρόνοιε στην Συμφωνία αποχώρηση για δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και δεύτερον την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Όσον αφορά το πρώτο, την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, φαίνεται να συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ότι η Ευρατόμ θα παραχωρήσει την ιδιοκτησία ε, ε, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που έχει και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα συνεχίσει να φροντίζει το Ηνωμένο Βασίλειο για την ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τα πυρηνικά απόβλητα, ε, θεωρείται ότι ότι το κράτος στο, το, στο οποίο παρήχθησαν θα πρέπει να είναι εκείνο το οποίο θα αναλάβει τον, ε, τη διαχείρισή τους. Τώρα, για το ζήτημα της, των επιπτώσεων στις, ε, της ενεργειακής ε, αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και, όσον αφορά τις εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι μετά τον Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα ακολουθεί τι ρυθμίσει, το ρυθμιστικό πλαίσιο τη ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και ότι θα ακολουθούνται οι αυστηροί κανόνες όσον αφορά την οικονομία, την, λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διαφάνεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσει κανείς την πιθανότητα να υπάρξει μείωση της αποτελεσματικότητας. Κατά την άποψή μας, θα συνεχίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι ένα σημαντικό κόμβο για το εμπόριο φυσικού αερίου. Ωστόσο, θεωρούμε ότι κάποιε ε, κόμβοι εμπορία φυσικού αερίου ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη ε, σημασία, γιατί πλέον αυτοί οι κόμβοι δεν θα, είναι δεν θα υπάρχει κίνδυνο συνδεδεμένο με τι διακυμάνσει του συναλλάγματο, όπω θα υπάρχει πια με την Ηνωμένο Βασίλειο. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιε άλλε περιοχέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία ω αποτέλεσμα του Brexit. Όπω έλεγα και στην αρχή, ένα ε, κρίσιμο ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι η επίπτωση τη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ιρλανδία και μάλιστα ένα από του άλλου συμμετέχοντε θα μιλήσει πιο συγκεκριμένα σε αυτό. Εδώ μπορεί να υπάρξουν σημαντικέ επιπτώσει. Γνωρίζουμε ότι η, ηλεκτρική, αγορά ηλεκτρική ενέργεια είναι ενιαία ε, μεταξύ τη δημοκρατία τη Ιρλανδίας και τη Βόρεια Ιρλανδίας και έχει σημαντικέ εισαγωγέ φυσικού αερίου 56% σα είπα προηγουμένω από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το καλύτερο ε, για την Ιρλανδία βεβαίως, θα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει ε, στην ε, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Η δεύτερη καλύτερη επιλογή θα ήταν η Βόρεια Ιρλανδία τουλάχιστον να παραμείνει στην ενιαία αγορά και η χειρότερη και τελευταία επιλογή θα ήταν τελικά να μείνει μόνο η δημοκρατία της Ιρλανδίας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού μετά το Brexit. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα χρειαστεί η Ιρλανδία αμέσως μετά το Brexit να της δοθεί κάποια παρέκκληση ώστε να μην ε, χρειάζεται να επιβάλλει ε, κάποιες από τις προβλέψεις των κανονισμών των ενεργειακών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως με δυσκολία μπορούμε να δούμε πώς θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η Ιρλανδία συνιστά πλέον ε, απομονωμένη ε, περιοχή ενεργειακά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Χρησιμοποιήσατε μόνο τα δύο τρίτα του χρόνου που είχατε στη διάθεσή σας, οπότε Περνάμε στον επόμενο ομιλητή μας, ε, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργ Σάχμαν και θα μας μιλήσει για τις επιλογές και τις σκέψεις για το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής ε, και της σύμπραξης για το αέριο με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Θα μας μιλήσει για όλα τα θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί, για την αλλαγή του κλίματος, γιατί έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής ε, Ρήπων, έχει ασχοληθεί με την αγορά των ε, προϊόντων, ε, με την συγκέντρωση της αγοράς, με την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Εκπομπών, το σχεδιασμό του συστήματος και με τις οικονομικές ε, επιπτώσεις στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, στη Μεσόγειο. Ε, είναι πολύ σημαντικό που και οι δυο σας ασχολείστε με τη Μεσόγειο και η συζήτησή μας γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο και Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόταση, για την πρόσκληση που μας δώσατε την δυνατότητα να έρθουμε εδώ. Μιλήσαμε για το θέμα. Σας έχω στείλει και ένα έγγραφο. Είναι 130 σελίδες και γι' αυτό θα προσπαθήσω να συνοψίσω σε 10 λεπτά το κομμάτι που αφορά στο ε, αέριο και την εμπορία αερίου εικόνα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι σχετικά καλού η εικόνα. Είναι βασικά χώρα ε, εισαγωγής αλλά και διαμετακόμισης προς την Ιρλανδία η Αγγλία. Είναι μια ενδιάμεση χώρα. Και το γεγονός ότι υπάρχει εμπόριο αερίου και με πολλές ε, μη ευρωπαϊκές χώρες ήδη και υπάρχει εμπειρία ε, μας δείχνει ότι θα μπορούμε να βρούμε μια αποτελεσματική λύση ε, πολύ και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα για την ανταλλαγή και την εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας το Ηνωμένο Βασίλειο και πάλι είναι βασικά εισαγωγέας. Αγοράζει ηλεκτρισμό από την υπηρετική Ευρώπη και συγκεκριμένα από τη Γαλλία και εξάγει στην Ιρλανδία. Το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχετικά περιορισμένο αν το συγκρίνουμε με το εμπόριο αερίου. Είναι μόνο 1,2 δις ή 10% του συνολικού όγκου του μέσου όγκου συναλλαγών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε το θέμα του συντονισμού όταν μιλάμε για τις αγορές ηλεκτρισμού, γιατί ο ηλεκτρισμός δεν είναι κάτι που μπορεί να αποθηκευτεί. Αν συμβεί κάτι στο Ηνωμένο Βασίλειο και ταυτόχρονα συμβεί κάτι στην Ολλανδία και στη Γαλλία, οπότε είναι σημαντικό να δούμε ακριβώς τι έχει στο μυαλό της Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανταλλαγές, εμπορικές συναλλαγές μάλλον σε εμπόριο για το μέλλον. Φαίνεται ότι θα αυξηθεί και γιατί είναι μεταβλητή αυτή η αγορά, αλλά και γιατί η δυνατότητα διασύνδεσης θα διπλασιαστεί του χρόνου και τα επόμενα έτη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, Ηνωμένου Βασιλείου γιατί θα είναι διαθέσιμες περισσότερες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκών και μη Ευρωπαϊκών χωρών, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη ε, ε χωρών που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εύκολο. Έχουμε δει ανταλλαγές με τη Μαρόκο, τη Φιλανδία και τις Βαλκανικές χώρες στο παρελθόν. Βέβαια δεν μιλάμε για ένα χίδιν εμπόρευμα το οποίο μπορείς να εμπορευθείς έτσι απλά, δεν μπορείς να εμπορευθείς κιλοβατόρες, αλλά ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η επιθυμία να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά ενέργειας. Υπάρχουν ε, διάφορες ροές ε, χρημάτων ε, προς διάφορες κατευθύνσεις, ε, συστήματα υποστήριξης για τα ανανεώσιμα μεταξύ διαφορών χωρών. Υπάρχει συντονισμός, ικανότητα συντονισμού και καλό θα ήταν να βρούμε έναν τρόπο να τα εναρμονίσουμε όλα αυτά έτσι ώστε να έχουμε αγορές ε, χοντρικής, εξισορρόπησης, επενδυτικών υπηρεσιών κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά πρέπει να αναπτυχθούν και αυτή η ανάπτυξη είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν ε, να δούμε ε, την Αγγλία εκτός αυτού του πακέτου. Όταν είσαι μέρος αυτού του πακέτου, ε, τότε μπορείς να είσαι και μέλος μια λειτουργικής αγοράς. Τι γίνεται μόνο όμως αν μια χώρα φύγει από αυτή την εσωτερική αγορά και πάει σε ένα, ε, σε ένα εμπόριο σαν αυτό που έχει η Ρωσία και το Μαρόκο της, ε, του τύπου του ΠΟΕ. Ας πούμε ότι υπάρχουν άνεμοι στη Βόρεια Θάλασσα και ενισχύουν τους αναμογεννήτρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό, ο ηλεκτρισμός δεν θα περάσει αυτόματα στην Ολλανδία, δεν υπάρχει πλέον ρευστότητα ε, στη συνολική αγορά, λιγότερος ανταγωνισμός, λιγότερα ωφέλη από αυτόν και αυτό που είναι το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε ε, λιγότερα σημάδια βέλτιστης ε, επένδυσης. Δηλαδή θα πρέπει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο να βρει τρόπο να χρηματοδοτήσει νέα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνάδουν με την υφιστάμενη αγορά και θα, μπορούμε στο τέλ, θα δούμε στο τέλος να έχουμε μια παραπάνω ε, παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο που δεν θα μπορεί να απορροφηθεί και το ίδιο θα γίνει και, στο, ε, και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτήν την καθαρά τομεακή ας πούμε οπτική γωνία ε, μια κοινή αγορά θα ήταν καλύτερη και για τις δύο πλευρές. Το να μείνουν τα πράγματα δηλαδή ως έχουν. Για να ξύσουμε λίγο την επιφάνεια και να δούμε από κάτω. Οι μηχανισμοί ικανότητα. αν βγει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, από την εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποφασίσει το ίδιο για την δική του τάση, για τη δική του ισχύ και δυναμικότητα. Ε, οι πελάτες λοιπόν θα πρέπει να έχουν αυτές τις επιλογές και η υπερβάλλουσα ισχύς η δυναμικότητα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα επενδύσεις ε, στην υπηρετική Ευρώπη ή στο Ηνωμένο Βασιλείο αντίστοιχα. Κάτι άλλο που ήδη αναφέρθηκε είναι ο, η αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών εταιριών στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία ως τώρα ήταν η πιο ανοιχτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό υπήρχαν μεγάλοι ε, παίχτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν επενδύσει εκεί. Ε, Scottish Power, E.ON, RWE Power. Άρα μετά από, την, ε, από το Brexit δεν θα έχουν ε, ας πούμε αυτές τις δεσμεύσεις ε, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα να είναι πιο δύσκολο οι εταιρείε αυτές να έχουν διακριτική μεταχείριση λόγω αυτών των αποφάσεων για τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης, άρα δεν θα είναι ίση η όρη. Επίσης, ποιο θα είναι το εύρος των ρυθμίσεων φαίνεται πως όλες οι συναλλαγές ε, πρέπει να... Ο Acer πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις συναλλαγές για να υπάρχει μια καλή παρακολούθηση της αγοράς και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίχτες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το εμπόριο πετρελαίου, ε, αερίου, αλλά και ηλεκτρισμού και εκπομπών. Τι γίνεται αν βγει εκτός του πεδίου των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν θα είναι πλέον δυνατή και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια διαφάνεια, να υπάρχουν κοινοί κανόνες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αλλιώς θα έχουμε μια ρυθμιστική μαύρη τρύπα. Όπως έχουμε δει και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μεγάλη η μάχη να μπουν αυτά τα, αυτές οι αγορές στο παιχνίδι. Για να συνοψίσω λοιπόν, από άποψη κλαδική και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ωφεληθούν αν μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει δεσμευμένο βάσει του κοινοτικού και εκτιμένου. Η κοινότητα ενέργειας και όχα είναι δύο διαφορετικά θεσμικά μοντέλα. Ε, βέβαια, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορούσε να είναι πλήρες μέλος της ε, κοινότητας της ενέργειας, αλλά υπάρχει το μοντέλο του ΕΟΧ. Υπάρχουν μοντέλα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Άλλες επιλογές επίσης ε, να είναι να πέσουμε τελείως στα στάνταρ του ΠΟΕ, δηλαδή ανταλλαγές χωρίς δασμούς ε, hidden ε, ποσοτήτων ηλεκτρισμού και αερίου, αλλά όχι τον ηλεκτρισμό στο επίπεδο που θα θέλαμε ώστε να έχουμε αποτελεσματική ενεργειακή αγορά. Η άλλη, ε, ε, αυτή η επιλογή επίσης ε, σημαίνει ότι θα είχαμε μια ένα σωρό λεπτομέρειες που θα έπρεπε να ρυθμιστούν σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα έπρεπε όλοι οι κανονισμοί και οι οδηγίες που σχετίζονται με την εμπόριο ηλεκτρισμού και αερίου να ξανά ε, ρυθμιστούν και αυτό θα ήταν μια τεράστια πρόκληση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τήρησατε και εσείς το χρόνο σας ευλαβητά, όπως όλοι οι μηχανικοί που σας έλεγα στην αρχή. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Διαπιστώνω ότι σε ένα μέρος της Ιρλανδίας ίσως να μην υπάρχει πρόβλημα. Αλλά η Ιρλανδία είναι δημιουργική ελληνικό και τι ξεπερνούν τι δυσκολίε. Και έτσι περνάμε λοιπόν στον, στην τρίτη ομιλήτρια, Λόρα η οποία θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις του Brexit στην ε, ενεργειακή αγορά της ε, Ιρλανδίας. Είναι διευθύντρια για ζητήματα αγορών ε, ενέργεια. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα της ενέργειας, της ενεργειακής πολιτικής, της τιμολόγησης σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Παλαιότερα έχει εργαστεί και ως σύμβουλος σε χρηματοοικονομικά θέματα και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντα συμβουλές σε ρυθμιστικές αρχές, σε κυβερνήσεις, σε ζητήματα όπως η ιδιωτικοποίηση και η τιμολόγηση, σε πολλέ χώρε ανάμεσα στις οποίες η Ταϊλάνδη, ο Καναδά, οι Ηνωμένε Πολιτείε και αλλού. Έχετε το λόγο κύριε Μπράιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κότσεκ και με ιδιαίτερο ευτυχή που θα έχω τη δυνατότητα σήμερα να σας μιλήσω για το εμπόριο της ηλεκτρικής ενέργειας και το ποιο θα είναι, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του Brexit σε αυτό. Ε, ακούστηκε ήδη το ζήτημα του φυσικού αερίου, η παρουσίασή μου όμως θα εστί στον ηλεκτρισμό. Να σας δώσω πρώτα απ' όλα κάποιες πληροφορίες για την ε, ΣΕΜ, την Κοινή Ενεργειακή Αγορά. Δημιουργήθηκε το 2007 ως μια αγορά χίδιν, η οποία καλύπτει τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη Βόρεια Ιρλανδία. Ε, συμμετέχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ιρλανδίας, στην οποία εργάζομαι, καθώς επίσης και η Ρυθμιστική Αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας. Η Επιτροπή ΣΕΜ δημιουργεί κοινού κανόνες για την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Και ε, υπάρχει ένα ε, σαφές νομοθετικό πλαίσιο και στις δύο χώρες που τη θεσπίζει. Ε, αυτό έχει οδηγήσει στο να έχουμε ένα κοινό ε, πλαίσιο κανόνων για όλους τους εμπορευόμενους, τους εμπλεκόμενους στην κοινή αυτή αγορά. Έχουμε ένα, ένα σύστημα για την αντιμετώπιση του γεγονότος ότι υπάρχουν δύο νομίσματα, το ευρώ και η στερλίνα, και ε, έχουμε δημιουργήσει ένα ε, σύστημα κοινό, συγχρονισμένο, για την διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ίσο της Ιρλανδίας. Η... Δημιουργήθηκε το 2007 ιστορικά αυτή η αγορά από Αργότερα βέβαια κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δημιουργήθηκε και η κοινή ευρωπαϊκή αγορά και το αντίστοιχο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επομένως επιδιώξαμε τη διασύνδεση με αυτήν. Αυτήν την στιγμή προσπαθούμε να ενισχύσουμε την διασύνδεση της κοινή ε, Ιρλανδικής αγοράς με την ευρωπαϊκή αγορά, όπως για παράδειγμα τις διδασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, την ε, εξισορρόπηση των φορτίων και διάφορα άλλα τέτοια θέματα. Προσπαθούμε να τα πράξουμε αυτά ε, για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των διασυνδέσεων και να αποτελέσουμε ένα, ε, μια αγορά η οποία συμμετέχει στην κοινή ενεργειακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα, ε, μπορεί να υποβάλει προσφορές για αυτήν την αγορά ως μια ενιαία αγορά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς κάποιους από την ε, Ευρώπη. Χρειάστηκε λοιπόν να δημιουργηθούν πολλές ε, διασυνδέσεις, μισό γιγαβάτ μεταξύ ε, Βόρειας Ιρλανδίας και Σκοτίας, μισό γιγαβάτ μεταξύ Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και Ουαλίας. Υπάρχουν επίσης και σχέδια για τη δημιουργία νέων διασυνδέσεων, πάλι μισό γιγαβάτ μεταξύ Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου αυτές οι διασυνδέσεις αντιπροσωπεύουν το περίπου 15% της ζήτησης, το οποίο είναι σημαντικό. Ε, αυτές οι διασυνδέσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της αγοράς της ε, ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία και επομένως είναι σημαντικό να έχουμε ε, αυτές τις διασυνδέσεις να λειτουργούν αποτελεσματικά γιατί μπορούμε να αξιοποιούμε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της υπόλοιπης Ευρώπης, της Ευρώπης. Μετά το Κατά τα άλλα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διασυνδέσεις περίπου 900... Ε, διάφορες διασυνδέσεις α, της τάξης του 1 γιγαβάτ με άλλες περιοχές της επιρωτική Ευρώπης και την Νορβηγία έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτει ε, τις ανάγκες του τις ενεργειακές σε περιόδους εχμής. Βεβαίως ε, κάποιες από αυτές τις διασυνδέσεις είναι παλαιές και ανακαινίζονται, κάποιες έχουν ξεκινήσει να ανασχεδιάζονται και κάποιες ήδη λειτουργούν. Ένα στοιχείο σημαντικό ε, της δικής μας αγοράς είναι ότι άλλαξε η μορφή του. Ιστορικά η κοινή Ιρλανδική αγορά είχε ξεκινήσει και να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 2016 στο 2017 αντιστράφηκε η τάση και εξήγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Ήθιστε να εισάγουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και να εξάγουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό επειδή έχουμε ε, μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ιρλανδία και έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το γεγονό ότι έχουμε ισχυρού ανέμους κατά την ε, νυχτερινή περίοδο ε, ε, και, βλέπετε στο γράφημα, που, αν το βλέπετε, ότι στις αρχές είχαμε σε μεγάλο βαθμό εισαγωγές μέσω των διασυνδέσεων, ενώ αργότερα περάσαμε σε καθαρές εξαγωγές ε, τα επόμενα έτη. Είναι σημαντικό να για την αποδοτικότητα του συστήματός μας να μπορούμε να, μετα... κάνουμε αυτή μετάπτωση από εισαγωγή σε εξαγωγή λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορές της τιμής. Λοιπόν, αυτή η κοινή αγορά Προφανώ δημιούργησε μεγάλες πλεονεκτήματα για την και η οικονομία και επιθυμούμε αυτό να συνεχιστεί και μετά το Brexit. Αυτό έχει βελτιώσει την ε, ε, ε, ενεργειακή μας ασφάλεια και έχει επιτρέψει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά συνολικά, αλλά και για τον Ιρλανδό καταναλωτή. Υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ε, ε, λύσουμε σε σχέση με το, ε, μετά το Brexit. Πρώτα απ' όλα είναι πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί η κοινή Ιρλανδική αγορά και δεύτερον ποιε θα είναι οι σχέσει οι εμπορικέ με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Γνωρίζουμε ότι το καλύτερο για εμάς θα ήταν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην, ενιαία, ε, στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Όμως φαίνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι να συνεχίσει να λειτουργεί η κοινή Ιρλανδική αγορά ενέργειας. Αυτό ε, είναι προτεραιότητα της Ιρλανδικής κυβέρνησης, το έχει δηλώσει και το κείμενο όσο έχει αυτή τη στιγμή στη Συμφωνία Αποχώρησης το κρίνουμε θετικά. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ε, ε, θα διευκολύνουν, ε, μάλλον κάνουν επιθυμητή τη συνέχιση της λειτουργία της κοινή ελληνικής αγοράς είναι το γεγονός ότι μια ευρωπαϊκή εταιρεία θα μπορούσε να κάνει προσφορές σε αυτή την αγορά ως ενιαία. Και επίσης διάφορα αλλαγέ στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα το πακέτο για την καθαρή ενέργεια, θα ενσωματώνονται. Εμείς επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο και οι κανόνες για τον ανταγωνισμό να είναι συμβατές με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωση όσον αφορά τις κρατικές ε, την εμπορία των ρήπων και το, το σύστημα για, αυτές, το, της συλλογής στατιστικών στοιχείων ή καθώς επίσης και την, ε, σημαντικό, το σημαντικό ρόλο που παίζει ο Acer στον συντονισμό των ρυθμιστικών αρχών των δικών μας με της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίλυση συγκρούσεων. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουν επίσης και οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο έτσι ώστε να γνωρίζουν ότι θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο δικαστήριο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν είτε αυτό είναι το, Ευρωπαϊκό, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε κάτι άλλο το οποίο θα συμφωνηθεί με την Συμφωνία Αποχώρησης. Το Brexit ε, όμως θα έχει επιπτώσεις και όσον αφορά την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ προσπαθούμε να, να φτιάξουμε κανονισμούς για να διευκολύνουμε την διασυνοριακή εμπορία ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μιας και η κοινή η Ιρλανδική αγορά είναι αυτή που είναι διασυνδεδεμένη άμεσα με το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την ευρωπαϊκή αγορά για πρόσβαση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η σε διαβούλευση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γνωρίζουμε ότι μετά τον Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο και οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται σε αυτό δεν θα έχουν πρόσβαση στι διάφορε πλατφόρμε για την εμπορία. Και για να, για να λυθούν αυτά τα προβλήματα θα χρειαστούμε κανόνες. Και προσπαθούμε να ε, εφαρμοστούν διμερώς οι κανόνες του, του ΚΑΚ που καλύπτονται σήμερα από αυτό και όσον αφορά τι τις ρυθμιστικές αρχές και όσον αφορά την εξέλιξη των διαφόρων συμφωνιών, πώς θα γίνουν οι συμφωνίες τώρα. Αυτές οι αλλαγές χρειάζονται χρόνο για να συμφωνηθούν και για να εφαρμοστούν. Επομένως για μας ε, σημαίνει αυτό ότι θα υπάρξει κόστος για τη, στη μεταβατική περίοδο χρειάζεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πολύ ενδιαφερόμενοι, πολύ εμπλεκόμενοι να συμφωνήσουν, αλλά επίσης να, να, να δημιουργηθούν και οι διάφοροι φορεί που θα διαχειρίζονται την διάδοχη κατάσταση. Και διαπιστώνουμε, πιστεύουμε ότι αυτές τις εμπορικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας με το Ηνωμένο Βασίλειο ε, θα πρέπει να τις δουν και πολλές άλλες χώρες, ενδιαφέρουν και πολλές άλλες χώρες πέραν της Ιρλανδίας δεν θα ήταν ε, ευκταίο να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου η Ιρλανδία θα κάνει διμερεί διαπραγματεύσει με το Ηνωμένο Βασίλειο για τα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν και άλλε χώρε οι οποίε ενδιαφέρονται, το Βέλγιο, οι κάτω χώρε, οι οποίε είτε έχουν διασύνδεση είτε ε, σχεδίαζαν να αποκτήσουν διασύνδεση. Επομένω, τι ενδιαφέρουν ε, αυτέ οι συμφωνίε μεταβατικέ. Επομένως αυτές οι διαπραγματεύσεις καλό θα είναι να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ και ερχόμαστε στην τελευταία ομιλήτρια που είναι η κυρία Μάλ, που θα μας μιλήσει για τον αντίκτυπο ε, της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στη Euratom. Εργάστηκε για την Φόρατομ από τον Ιούνιο του 2004 και έκτοτε έχει αναλάβει την διαχείριση και τον παροπλισμό πυρηνικών υλικού και έχει ασχοληθεί και με νέα πυρηνικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είναι υπεύθυνη για την ανάλυση των επιπτώσεων του Brexit όσον αφορά την πυρηνική βιομηχανία. Έχετε το λόγο κυρία Πικαμάλ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πράγματι, στην πυρηνική βιομηχανία ε, υποκείμεθα στην ε, Συμφωνία Euratom και από τη στιγμή που θα αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο αρχίσαμε να αναλύουμε και εμείς τις επιπτώσεις για την Ευρώπη των 27 από την αποχώρηση αυτή και θα σας παρουσιάσω κάποια συμπεράσματα στο οποία καταλήξαμε. Για όσους δεν γνωρίζετε την ΦΟΡΑΤΟΜ, είμαστε ένας οργανισμός της πυρηνικής βιομηχανίας της Βρυξέλλες. Οπότε έχουμε επαφές με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλους τους ενδιαφερόμενους. πόσο συνεισφέρει η πυρηνική βιομηχανία στην ευρωπαϊκή οικονομία σήμερα. Υπάρχουν 127 πυρηνικοί σταθμοί, αντιδραστήρες μάλλον, στις 28 χώρε, δηλαδή και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για 70 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο ε, που στηρίζουν πάνω από 800.000 θέσεις απασχόλησης. Και η πυρηνική ενέργεια προσφέρει το 27% του ηλεκτρισμού, της ηλεκτρικής παραγωγής. Τώρα, ποιο είναι καταμερισμό στι διάφορε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά του πυρηνικού αντιδραστήρε που έχουμε στο έδαφο μα. Και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλω να σα δείξω σήμερα είναι αυτό. Δηλαδή, ποια είναι τα σχέδια οικοδόμηση. Και θα δείτε στο χάρτη ότι υπάρχουν πολλά σχέδια ε, για πυρηνικούς ε, αντιδραστήρες στο Ενωμένο Βασίλειο στο μέλλον. Και μιλάμε για 68 δισεκατομμύρια ευρώ. Για παράδειγμα, το 1 τρίτο της αξίας οικοδόμησης ενός από το πιο γνωστού του HPC αντιδραστήρα ε, θα προέλθει από την Ευρώπη των 27. Πάνω από 5 δισεκατομμύρια ε, συμβάσεις έχουν, ε, για τέτοια ποσά δηλαδή συμβάσεις έχουν υπογραφεί με την Ευρώπη των 27. Οι πυρηνικοί σταθμοί όταν λειτουργούν όμως χρειάζονται και συντήρηση. Και τα νούμερα που θα σας δώσω τώρα δεν συμπεριλαμβάνουν τα καύσιμα ή τα επιπλέον συστατικά Πρόκειται για τη λειτουργία, τη συντήρηση των μονάδων που ήδη υπάρχουν, που είναι αξία 48 εκατομμυρίων κατέτος. Και τα χρήματα πάνε και σε επιχειρήσεις της Ευρώπης των 27 βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπογραμμίσουμε ότι όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, Υπάρχει ένας προπολογισμός παροπλισμού ετήσιος 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ που θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο από τα μέσα του 2020 γιατί θα αρχίσει να κλείνουν σταθμοί. Αυτό δείχνει γιατί νούμερα μιλάμε όταν μιλάμε για την πυρηνική ενέργεια και για το πόσο μπορεί να επηρεαστεί η πυρηνική βιομηχανία στις υπόλοιπες χώρες μέλη μετά το Brexit. Πριν από μερικούς μήνες αρχίσαμε να αναλύουμε πραγματικά τα νούμερα ε, από τις συνέπειες του Brexit στην πυρηνική βιομηχανία. Όντας μέσα και στο γεωροτομικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθήσε τους ίδιους κανόνες για την ασφάλεια. Τώρα, εκτός EuroTOM, αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διαπραγματευτεί ένα καθεστώς με την ε, Διεθνή Υπηρεσία Πυρηνικών που θα είναι αντίστοιχη με αυτή που έχουμε σήμερα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξακολουθεί να έχει σχέσεις με την πυρηνική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου με νέες συμφωνίες βέβαια μετά το Brexit που τους ονομάζουμε NCAs. Υπάρχουν τέτοιε συμφωνίες με άλλες τρίτες χώρες, οπότε το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον θα γίνει τρίτη χώρα, θα πρέπει να υπάρχει τέτοια συμφωνία NCA και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης υπογραμμίζουμε και τη σημασία που έχει η εγκυρότητα των ε, συμβάσεων. Υπάρχουν συμβάσει που έχουν υπογραφεί πριν από το Brexit και που ε, θα πρέπει μετά από το Brexit να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει με αυτές. Πρέπει να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι αυτές οι συμβάσεις θα εξακολουθούν να είναι έγκυρες ακόμα και μετά το Brexit. Παρά το γεγονός ότι η πυρηνική βιομηχανία ε, ακολουθεί τη συνθήκη Euratom, ε, εμπίπτουν σε αυτό και θέματα ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και θέματα εσωτερικής αγοράς. Είμαστε ένα συνολικός κλάδος. Η κυκλοφορία ατόμων λοιπόν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο πάντα διευκολύνεται και διασφαλίζεται. Και θα θέλαμε να συνεχιστεί αυτό. Όσον αφορά τώρα τα άλλα τετραγωνάκια που βλέπετε εδώ, R&D, έρευνα και ανάπτυξη, υπάρχει ένα πρόγραμμα από τον προπολογισμό της Euratom στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Κόλομ, οπότε Οπότε η έρευνα αυτή συνεισφέρει στο ΙΤΕΡ που είναι ένα διεθνέ πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξουν κάποια στιγμή σε συμφωνία για το πώ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στην έρευνα και την ανάπτυξη. Για να μην ε, σταματήσουν ή ενοχληθούν, εν πάση περιπτώσει, τα προγράμματα τα διεθνή, τα οποία έχουν σήμερα από κοινού. Σημασία έχει και η στενή σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να παίζει ρόλο σε οργανισμούς όπως είναι το ΕΝΤΡΑΚ. Έχοντας αναλύσει τώρα τις συνέπειες για την πυρηνική βιομηχανία μετά το Brexit, ένα από τα ζητήματα τα οποία είναι πιο προφανή είναι το εξή τι θα γίνει με τις αρχές, τις βασικές αρχές που θέλουμε να αναπτυχθούν σε μελλοντικές σχέσεις ανάμεσα στην Euratom και το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω συμφωνίας NCA για παράδειγμα που σας έλεγα και πριν. Πολλές αρχές βέβαια υπάρχουν, αλλά εδώ αναφέρω πέντε που είναι οι πιο σημαντικές. Ελεύθερο εμπόριο για υλικό πυρηνικό και μη πυρηνικό να διασφαλίσουμε δηλαδή το ελεύθερο ε, εμπόριο για τέτοια αγαθά και υπηρεσίε. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζόμενων ε, στον πυρηνικό κλάδο. Όπως είπα και πριν, έτσι κι πρόκειται για έναν πανευρωπαϊκό κλάδο. Οπότε έχει μεγάλη σημασία η ελεύθερη κυκλοφορία για μας. Έπειτα, άλλο σημαντικό είναι η έγκριση των ε, συμβάσεων που έχουν υπογραφεί νωρίτερα, πριν από το δημοψήφισμα δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να διασφαλιστεί η εγκυρότητά τους και στο μέλλον. Έπειτα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι ακριβώς οι επιπτώσεις από τον έλεγχο των εξαγωγών και τις σχετικές άδειες. Και βεβαίως πρέπει τέλος να διασφαλίσουμε τη διεθνή συνεργασία να παραμείνει στα θέματα έρευνας και ανάπτυξης στον πυρηνικό κλάδο. Ευχαριστώ. Και κάτι ακόμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό το οποίο αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς από τη δική μας την πλευρά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές ασφάλειας της IAEA. και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει προδιαγραφές για την ε, προστασία ε, κάθε φορά που υπάρχει μεταφορά υλικού, μαγαθών, εξοπλισμού κτλ. Οπότε για να έρθω στην αρχή των παρουσιάσεων σώσα να φέρε Σιμώνε για τα πυρηνικά Πράγματι υπάρχουν δύο ζητήματα που θεωρούμε τα πιο σημαντικά. Η ασφάλεια, και εσείς το είπατε, και άλλο είναι η ασφάλεια και άλλο είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες για μας. Και το δεύτερο είναι το θέμα των αποβλήτων. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις, για τα δύο ζητήματα, Υπάρχουν συνολικές συμφωνίες με κάποια συμπεράσματα, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε πιο συγκεκριμένα στις επιπτώσεις στην οικονομία των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ευχαριστούμε πολύ και σας. Τηρήσατε το χρόνο σας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπάρχει η δυνατότητα, όποιος ενδιαφέρεται από τα μέλη της Επιτροπής μας, να παρουσιάσει τις ιδέες του και φυσικά να κάνει και ερωτήσεις. Μια που σας έχουμε εδώ. Και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Κέλλη είναι ο πρώτος συνάδελφος, η κυρία Φαν Μπρέμπτ είναι η δεύτερη, ο κύριος Φλοκ. Ωραία. Θα ακούσουμε μερικές ερωτήσεις και μετά θα σας δείσουμε να απαντήσετε. Ωραία, αρχίζουμε λοιπόν. Παρακαλώ κύριε Κέλλη, εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας. Γιατί παρουσίασαν μια κατάσταση που θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ περίπλοκη, με απλά λόγια. Μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε και ακούσαμε και τα συμπεράσματα. Είμαι ο μόνος Ιρλανδός εδώ στην Επιτροπή αυτή βιομηχανία. οπότε σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Για μας, για την Ιρλανδία, τη χώρα μου, είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό. Όταν μιλάμε για τις συνέπειες του Brexit, είναι από τα κύρια ζητήματα αυτό. Βλέπετε και από τις παρουσιάσεις ότι για το φυσικό αέριο 56% φτάνει σε εμά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αν κάτι πάει στραβά, αν για παράδειγμα υπήρξε αδυναμία εφοδιασμού, γιατί δεν υπήρχε αρκετό φυσικό αέριο για την υπόλοιπη Ευρώπη, ε, θα είμαστε οι πρώτοι που θα υποφέρουν. Έχει βέβαια νόημα αυτό που λέμε ότι το καλύτερο θα ήταν να παραμείνει στο ΑΙΕΜ το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά αυτό που κολλάει με τόσο είχε πει ο κύριος Μπαρνιέ ότι δεν θα υπάρξει επιλεκτικό Brexit, δηλαδή σε άλλα ναι, σε άλλα όχι. Πώς δηλαδή ταιριάζει αυτό. υπάρχουν αυτοί που θέλουν το hard Brexit. Οπότε πού κολλάει αυτό σε σχέση με τις επιθυμίες αλλά και υποχρεώσεις που έχει ο κύριος Μπαρνιέ να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει αυτό το επιλεκτικό Brexit. Θα ήθελα τις απόψεις σας από αυτού. Και κάτι ακόμα για τις διασυνδέσεις Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Μια γενική ερώτηση έχω. Σε ποιον ανήκουν οι διασυνδέσεις αυτές. Και αν υπήρξε σκληρό Brexit, ποιος θα είναι υπεύθυνο, τι θα γίνει με αυτούς, θα κλείσουν, θα διατηρηθούν. Και αν δεν είναι το Ηνωμένο Βασίλειο στον ΑΙΕΜ. Πάντα για την Ιρλανδία. Θα συμφωνήσει και η Λάουρα δίχως άλλο. σύνδεση Ιρλανδίας-Γαλλίας. Αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία σήμερα δεδομένου του Brexit. Γιατί αν μη τι άλλο θα είχαμε έναν interconnector με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Γαλλίας. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τη γνώμη σας. Και πείτε μου που να σταματήσω, ε, γιατί θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες. Σε σχέση με την ε, ενιαία αγορά ενέργειας, τι δεσμεύσεις αναλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με το backstop, αν ε, δηλαδή ακολουθήσουμε αυτές τις λύσεις έκτακτης ανάγκης που λέμε. Και τέλος για τα πυρηνικά. Δεν έχουμε πυρηνικά στην Ιρλανδία. Αναφέρεστε στα πυρηνικά στην Ευρώπη, στους πυρηνικούς σταθμούς στην Ευρώπη. Πόσοι από αυτούς τους ε, σταθμούς βρίσκονται στο Ενωμένο Βασίλειο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί δεν βλέπω τα νούμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, υπομονή σας αλλά επειδή είμαι ο μόνος Ιρλανδός εδώ, ήθελα να τα έχω πει αυτά και σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρουσιάσεις σας. Σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά σας. Ε, ξεπεράσατε λίγο τον ε, χρόνο σας, 150% που σημαίνει ότι είστε πραγματικός πολιτικός. Ευχαριστώ η κυρία Φαν Μπρέντ, έχει το λόγο. Πόση ώρα έχω. Δύο λεπτά. Ωραία. Νομίζω ότι ο κύριο Κέλλη έχει κάθε δικαίωμα να ανησυχεί γιατί το θέμα αυτό πραγματικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ευχαριστώ. Έμαθα πολλά. Πολλά από αυτά τα ζητήματα δεν τα είχα λάβει καν υπόψη μου. Έχω ένα πιο γενικό ερώτημα. Όσον αφορά στην εσωτερική αγορά, νομίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος να το εντομετωπίσουμε είναι να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ενεργειακή Ένωση, να πάρει μαζί του όλο το κεκτημένο και για το μέλλον, όχι μόνο για τα τεχνικά στοιχεία και τα στοιχεία της αγοράς, αλλά και για την κοινή δράση που έχουμε ως προς την ε, βιωσιμότητα κτλ. Και αυτό είναι και το ερώτημά μου βασικά. Αν δούμε το πιο μακροπρόθεσμο μέλλον και τις δεσμεύσεις που έχουμε όλοι μας. Κάποια στιγμή θεωρώ ε, νωρίς ή αργά θα πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα με πλήρη ε, τροφοδότηση από τα ανανεώσιμα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η σύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και υπόλοιπη Ευρώπης δεν είναι τόσο μεγάλο ε, πρόβλημα τώρα, αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο, αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί. Εκτός αν μου πείτε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο μπει στο η γραμμή αυτή για την ε, αποδοτικότητα πλήρως με ΑΠΕ ε, χωρίς να βοηθά η Ευρώπη. Έχετε κάποια νούμερα γι' αυτά, θα με ενδιαφέρε πολύ. Και κάτι πιο πολιτικό ως σχόλιο σχετικά με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Επειδή από ό,τι διάβασα δεν υπάρχει πρόθεση να παραμείνουν στην Ενεργειακή Ένωση, ως τώρα τουλάχιστον, αυτό λέει στη Λευκή Βίβλο, θεωρώ ότι στις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή για την αποδοτικότητα και τα ανανεώσιμες, βλέπουμε ένα τεράστιο λόμπι από το Ηνωμένο Βασίλειο που προσπαθεί να εξασθενήσει αυτή τη θέση, κάτι που για μένα φαίνεται περίεργο. Είναι πολιτικό το ερώτημα αυτό, αν έχετε όμως κάποιες πληροφορίες ή μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο, δεδομένου ότι θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι συμφέρον έχει να εξασθενήσει κάπως ε, τις, ε, την νομοθεσία σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ανανεώσιμες κλπ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Ο κύριος Μπούλοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις. Ε, με χαρά μου βλέπω ότι σύμφωνα με τον ΠΟΕ μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να εισάγει και να εξάγει ενέργεια χωρίς ε, δασμούς ε, σε άλλες χώρες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά αν και αλλά στις παρουσιάσεις και διάφορες πιθανότητες και δυνατότητες όταν κρίνουμε το τι ενδεχομένως να συμβεί. Ε, αυτό ακριβώς συνέβη και σε όλη τη διαδικασία και την εκστρατεία για το δημοψήφισμα. Τελικά, ε, από όλα αυτά τα σενάρια έχει το Ηνωμένο Βασίλειο ε, έλεγχο για τις υποθέσεις του. Αυτό ίσως είναι το σενάριο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν όχι, ε, τότε ε, τι θα γίνει αν φύγει. Έτσι πρέπει να σκεφτούμε νομίζω. Κάτι άλλο, ας πούμε ένας τρόπος να ανακτήσει τον έλεγχο είναι στο μέλλον να μειώσει διάφορους φόρους, ας πούμε τον ΦΠΑ για την ενέργεια, για τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο. Αν γίνει αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βόρεια Ιρλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία γενικά, τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην νήσο της Ιρλανδίας, στην νήσο Ιρλανδία. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε το νούμερο ένα ως προς την τήρηση του χρόνου. Και τώρα η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Και εγώ θα είμαι σύντομη στο χρόνο σίγουρα. Έχω μόνο μία ερώτηση και η παρατήρησή μου είναι ε, ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις εκτενείς και πολύ συγκεκριμένες ε, και ενημερωτικές ε, παρουσιάσεις τους μας έθεσαν όλα τα επίπεδα της πολιτικής για το Brexit. Οι τέσσερις αυτές ε, παρουσιάσεις, αν τις αξιολογήσω, βγάζω το συμπέρασμα ότι με την εξαίρεση της Ιρλανδίας εμείς δεν θα έχουμε προβλήματα μετά από το Brexit στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική. Μπορούμε να τα λύσουμε όλα με τάξη και ασφάλεια. Και για το σύστημα ETS ε, και για την ε, Συμφωνία του Παρισίου και για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο. Ε, αν λάβω υπόψη λοιπόν τα όσα είπατε, Ε, θα με ενδιέφερε να μάθω ακόμα ε, αν σε ερευνητικό επίπεδο υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το πώς ε, θα διαμορφωθούν τα πράγματα αν γίνει ένα φιλικό διαζύγιο και έχουμε στο μέλλον μια σύμπραξη. Σίγουρα Βέβαια, για το θέμα της Ιρλανδίας δεν λύνονται όλα τα προβλήματα, το είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και ένας άλλος τομέας. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε μια λαμπρή εξαίρεση μαζί με τον κύριο Μπούλοκ ως προς την τήρηση του χρόνου. Και τώρα έχω και πολλά απλά ερωτήματα που θα ήθελα εγώ να θέσω γιατί είμαι αυτός που προεδρεύει. Αλλά, εκτός από αυτό, είμαι και εγώ ευρωβουλευτής. Τι γίνεται με τους ε, επιστημονικούς αντιδραστήρες. Υπάρχει μια μεγάλη ε, συνεργασία, ε, ακόμα και στη Βιέννη υπάρχει ένα κάτι τέτοιο δίπλα στο Πανεπιστήμιο, στην Πράγα εκεί άλλα δύο και φυσικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία. Τι γίνεται με αυτόν τον τομέα γιατί είναι κάτι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο για τον ενεργειακό τομέα αλλά για τις εφαρμοκές. Ε, βλέπουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό νέων εφαρμογών, ας πούμε, στην ιατρική, στη βιομηχανία. Τι γίνεται με αυτή τη συνεργασία, σε αυτόν τον τομέα. Μετά, άνθρακας και κόκ. Τι γίνεται με το ισοζύγιο στην Βρετανία επηρεάζεται αυτό. Είναι βιομηχανική χρήση και είναι πολύ σημαντικό. Επίσης Εμονά και μάνατζερ ε, διευθυντής ε, σε ένα εργοστάσιο χάλιβα και το ξέρω και αυτό. Επίσης ε, το πετρέλαιο. Μιλήσαμε για ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο. Τι γίνεται με το πετρέλαιο. Και τέλος. Τι γίνεται με τα αποθέματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει τέτοια αποθέματα η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί ε, όλα τα κράτη πρέπει να έχουν τριών μηνών απόθεμα σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Ωραία. Θα πρότεινα να σας δώσω το λόγο, να δώσω το λόγο στους ομιλητές του πάνελ με την ίδια σειρά με την οποία κάνατε τις παρουσιάσεις σας αρχικά για να απαντήσετε. Επομένω ξεκινούμε από τον κύριο Τελιαπέτρα και με τους υπόλοιπους ομιλητές κατόπιν. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα απαντήσω στις ερωτήσεις που σχετίζονται με τη δική μου παρουσίαση, ξεκινώντας από αυτό που ρώτησε η κυρία Φαμπρέντ και την ερώτησή σας για τη διασύνδεση. Οι διασυνδέσεις είναι ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να δώσει ευελιξία στο σύστημα και ε, να κάνει το σύστημα ε, ικανό να υποδεχτεί όλο και περισσότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών. Θα έλεγα λοιπόν ότι το Brexit δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την εγκατάλειψη της χρήσης του, του άνθρακα στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί η διασύνδεση είναι μία από τις μεθόδους, υπάρχουν επίσης και άλλες μέθοδοι όπως η αποθήκευση όπως σωστά είπατε, επομένως δεν προβλέπεται ότι θα σταματήσει, θα, θα υπάρξει πρόβλημα με την ε, ε, εγκατάλειψη της χρήσης του άρθρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι οι τρέχουσες διασυνδέσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν, θα βρεθεί ένας τρόπος να συμφωνηθεί, ε, ένας τρόπος να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτές οι υποδομές. Κατά την άποψή μας, δεν υπάρχει λοιπόν κίνδυνο στο Brexit να σταματήσει αυτή είναι η διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να απαντήσω στην κυρία Νίμπλα, βασικά απάντηση είναι ναι. Έχετε δίκιο. Η μελέτη μας κατέδειξε ότι χρειάζεται να βρεθεί ένας τρόπος για τη διαχείριση, μάλλον θα βρεθεί ένας τρόπος για να διαχειριστούμε όλα τα θέματα εύκολα. Ε, το μόνο διζήτημα είναι η Ιρλανδία. Όπως σωστά είπατε και εσείς. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό, για αυτό που με ρωτήσατε για το, τον άνθρακα και το κόκ. Δεν ζητήθηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας να σταθούμε σε αυτά τα δυο στοιχεία του, του, του ενέργεια, της ενέργειας. Εμείς εστιάσαμε στον ηλεκτρισμό και το φυσικό ε, ε, αέριο. Και για έναν βασικό λόγο, η αγορά άνθρακα είναι μια παγκόσμια αγορά. Εξαιτία της, της φυσικής για την μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας χρειάζονται ε, εγκαταστάσεις αγωγή και αγωγή για την μεταφορά του φυσικού ε, αερίου. Ενώ για την εμπορία άνθρακα δεν βλέπω πώς το Brexit θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε αυτή την αγορά. Ε, και το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο. Ε, συγγνώμη, το, το πετρέλαιο. Επομένως, ούτε το πετρέλαιο ούτε ο άνθρακας θα επηρεαστούν από το Brexit συγκεκριμένα. Γι' αυτό και εστιάζουμε τη συζήτησή μας στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο. Να απαντήσω κι εγώ με τη σειρά μου. Αυτά που ρώτησε ο κύριο Σκέλη, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι δεν μπορεί να υπάρχει επιλεκτικό Brexit, δηλαδή να πάρει ό,τι θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο και ότι δεν θέλει να το αφήσει. Τώρα όμω ε, πρόκειται για cherry picking ή είναι κάτι από το οποίο έχουν εξυπηρετηθούν και οι δύο πλευρές. Αυτό πρέπει να το δούμε με την ενεργειακή κοινότητα. Κατά πόσο δηλαδή θα επιτραπεί τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει στη Eurotom και βέβαια να δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις. Έτσι θα παρέμενε άθικτη η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Κατά τα άλλα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μόνο να κερδίσουν έχουν ε, από συνεργασία μεταξύ τους. Και για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ζωτική σημασίας η Ιρλανδία να παραμείνει στο ενεργειακό σύστημα. Αλλιώς πώς θα λειτουργήσει ανεξάρτητα το σύστημα του, της Βόρειας Ιρλανδίας αν δεν υπάρχει διασύνδεση με την υπόλοιπη δημοκρατία. Γι' αυτό ρώτησε ο κύριος Μπούλοκ τώρα για το κόκ. Ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο, η ενέργεια δεν είναι συνηθισμένα αγαθά τα οποία εμπορευόμαστε στον ΠΟΕ. Πρόκειται για υπηρεσίες χρειάζονται υποδομές και χρειάζονται και θεσμοί οι οποίοι να διασφαλίζουν ότι ο αέρας φυσάει στη μια χώρα αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει σε κάποια άλλη και αυτό να λαμβάνεται υπόψη. Οι επενδύσεις είναι σημαντικό να γίνονται και από τις δύο πλευρές. Οπότε στο θεσμικό, το θεσμικό μας πλαίσιο βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν βλέπω αλλιώς να υπάρχει εμπόριο ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να επαναλάβω αυτό που είπε και η Σιμώνα, σε απάντηση στην κυρία Νίμπλερ, νομίζω ότι καλά συνοψίσατε βλέπουμε ότι η Ιρλανδική περίπτωση είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο, όπως λέμε, που θα πρέπει να λυθεί. Τα άλλα είναι πολύ λεπτομερή, μικρά ζητήματα. Τα νούμερα, η ρύθμιση, δημοσιονομικοί κανονισμοί, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς πού κρύβονται τα προβλήματα και πώς θα εμφανιστούν ε, πού και πότε. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για να φτιαχτεί μια νέα σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανταλλαγή ενέργειας με ναι, συμβάσεις, συμφωνίες, ρυθμίσεις. Αλλά άλλο ζήτημα τόσο κρίσιμο όσο το Ιρλανδικό δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Πράιεν. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Για να απαντήσω σε ερωτήσεις του κύριου Κέλλη πρώτα απ' όλα. Πράγματι υπάρχει μια έκθεση σκοπιμότητας που ετοιμάζεται ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιρλανδία από τους φορείς συστημάτων διασύνδεσης των χωρών αυτών. Και από πλευρά της Ιρλανδίας βλέπουμε να μπορεί να επωφεληθεί όχι τόσο πολύ από την ασφάλεια σίγουρα, εμείς χαιρόμαστε να υπάρχει μια, ένα ολοκληρωμένο σύστημα με κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα προφανώς και σίγουρα θα βοηθούσε πολύ την ολοκλήρωση της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πολλά ωφέλη για μας. Αλλά και όσον αφορά τις ε, τιμές ενέργειας. Η ολοκλήρωση με μια άλλη χώρα που έχει ένα διαφορετικό ενεργειακό μείγμα σίγουρα μας δίνει περισσότερες δυνατότητες εισαγωγών-εξαγωγών και σύγκριση τιμών Γαλλίας-Ιρλανδίας. Θέλουμε μια τέτοια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για τους διασυνδετήρες αγωγούς. Υπάρχει ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Ουαλία. Υπάρχει το Ιρλανδικό σύστημα λειτουργίας. Υπάρχει και ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκοτία που ανήκει σε μια μηδέα εταιρεία, πρόκειται δηλαδή για μια ιδιωτική επένδυση και υπάρχει επίσης ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα δεν θυμάμαι 100% Νομίζω ότι και εκεί πρόκειται για ιδιωτική επένδυση. Για τη ρύθμιση τώρα, τη συντήρηση κλπ. Η ρύθμιση γίνεται συνήθως από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οπότε η ΕΚ, ο διασυνδετικός αυτός αγωγός, έχει άδεια με υποχρεώσεις συμμόρφωσης Και το ίδιο ισχύει και ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, που τη λειτουργία τους λαμβάνει πολλές φορές ανάλογα, μπορεί η Γερμανία, μπορεί η Γαλλία. Αυτό που μας απασχολεί πιο πολύ όσον αφορά το εμπορικό σκέλος, πώς ο κόσμος θα έχει πρόσβαση στους αγωγούς αυτούς. Αν δηλαδή η παραγωγή γίνεται στη Γαλλία και εμείς ε, θέλουμε να έχουμε πρόσβαση από μια άλλη χώρα, πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση. Είναι θέμα της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οπότε αν το Ηνωμένο Βασίλειο βγει από αυτήν την αγορά, τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος διακανονισμός. Για να μην απομακρυνθούμε πολύ από την αποτελεσματική λύση που έχουμε τώρα. Και όσον αφορά τη συνέχεια... του ΣΕΜ στην Ιρλανδία. Εμείς ελπίζουμε ότι η νέα συμφωνία θα καταλήξει κάπου, θα μπουν υπογραφές. Και το παράρτημα 2.7 είναι το σημείο όπου συγκεκριμένα στοιχεία του τι χρειάζεται να εφαρμοστεί στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ιρλανδία για να παραμείνει το ΣΕΜ. Εκεί πρέπει να αναφερθούν. Οπότε ελπίζουμε το παράρτημα αυτό να διατυπωθεί όπως πρέπει. Και για τις άλλες ερωτήσεις ο κύριος Μπούλκ νομίζω ρώτησε. Για το ΒΑΣ. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό έχει να κάνει με τους λογαριασμούς λιανικής πώλησης. Δεν βλέπουμε να πρόκειται για θέμη το ανταγωνισμό, για το ΦΠΑ δηλαδή. Η παραγωγή τις δύο πλευρές της Ιρλανδίας δεν θα βρεθούν σε ανταγωνισμό, ελπίζουμε. Αν υπάρχει κάποια διαφορά ε, φορολογική, δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει τα πράγματα. Δεν, ξέρω, δεν είναι και ο τομέας μου ακριβώς. Πάντως αν υπάρχει αλλαγή, προφανώς θα υπάρξει αλλαγή και στις συνθήκες ανταγωνισμού. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ και τέλος η κυρία Πίκα Μάλ. Ναι, και εγώ να απαντήσω στις ερωτήσεις. Στον κύριο Κέλλη πρώτα απ' όλα. Θα σας στείλω τις διαφάνειες αν θέλετε. Υπάρχει η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα. Με έναν δύο αντιδραστήρες η καθεμία που σχεδιάζονται τώρα. Είναι Βουλγαρία, η Τσεχία, η Φιλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο για παραπάνω προγράμματα από αυτά που έχουν ήδη ξεκινήσει. Υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό. Ίσως να το έχετε ακούσει. Υπάρχει και το Sizewell, το Wilfer, στην Ουαλία επίσης. Υπάρχουν δηλαδή σχέδια, είτε υπό οικοδόμηση, είτε απλώ ε, στα χαρτιά. Για την έρευνα και τους αντιδραστήρες. Είκοσι περίπου ερευνητικοί αντιδραστήρες υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη και σε πυρηνικές χώρες και σε μη πυρηνικέ. Έτσι και αυτές έχουν τέτοιους αντιδραστήρες. Για μας είναι σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την έρευνα και την ανάπτυξη. Μπορούμε να εμπνευστούμε από πρόσφατες συμφωνίες με την Ουκρανία ή την Ελβετία, για παράδειγμα, που είναι συνδεδεμένη χώρα. Άπαξ και αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα υποφελείται πια από το Horizon 2020 ή άλλα ερευνητικά προγράμματα. Όπως είπατε, δεν πρόκειται μόνο για τον ηλεκτρισμό, πρόκειται και για τις συντήσεις, για εφαρμογές στη βιομηχανία κλπ. κλπ. ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι πιστεύουμε ότι το Horizon 2020 θα έπρεπε να είναι ανοιχτό και για άλλες χώρες, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχε γίνει μέχρι τώρα, αν μπορούν να συμμετέχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί όχι το Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύω ότι θα λυθούν αυτά τα προβλήματα στη βιομηχανία. Άλλα είναι τα θέματα διαπραγματεύσεων βέβαια. Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτό που κάνει είναι ότι περιγράφει την κατάσταση με ένα μεγάλο ερωτηματικό γύρω από την Ιρλανδία. Αυτό είναι πολύ βασικό και για τις δύο πλευρές που διαπραγματεύονται. Ήταν πλούσια η συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ε, προσκεκλημένους μας και ομιλητές μας εδώ. ladies and gentlemen, Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι χαρά που βλέπω ε, τον κύριο Μπουτούσνικ για άλλη μια φορά στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμά θυμάμαστε τις συζητήσεις μαζί του. Ήταν πάντοτε εξαιρετικές. As well as Mr. Ο, ο εκτός από τον κύριο Ποτότσνικ έχουμε και τον κύριο ε, που είναι ο πρόεδρος ε, του Συμβουλίου του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, ACER. Ανταλλαγή απόψεων με τον Άσερ είναι το όνομα αυτής της ε, ε συζήτησης που θα κάνουμε τώρα. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις? Όχι. Να σας θυμίσω ότι ο Άσερ προσεκλήθη για να μας δώσει μια ενημέρωση σχετικά με την δουλειά, την πρόοδο και τις ε, διάφορες προκλήσεις που παραμένουν για την ολοκλήρωση της αγοράς. Ε, μιλάμε για ένα αριθμιστικό ε, πλαίσιο, για το πακέτο ε, για την πράσινη ενέργεια και γενικά για τις δραστηριότητες του οργανισμού. Τέλος, ε, θα μας δώσουν και κάποια στοιχεία για τη δημοσιονομική κατάσταση του οργανισμού, αλλά και ε, κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τις οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, διότι αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε μια συζήτηση για το μέλλον, για τη μελλοντική δημοσιονομική περίοδο. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας και στις 5 η ώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να μπούμε αμέσως στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Γκάρετ και εγώ Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε για άλλη μια φορά να μιλήσουμε στην Επιτροπή σας. Θα σας κάνουμε μια μικρή παρουσίαση και μετά είμαι έτοιμος για ερωτήσεις και σχόλια. Η παρουσίαση μου επικεντρώνεται στις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Έχουμε κάποια καλά νέα να σας πούμε, αλλά θα σας μιλήσουμε και για τις πρόσφατες δραστηριότητες και τις προκλήσεις. Και μάλλον αυτές θα τις γνωρίζετε, τις προκλήσεις, γιατί είναι μπροστά μας εδώ και πολύ καιρό. Χωρίς άλλη λοιπόν καθυστέρηση, περνάμε στην παρουσίαση. Μπορεί να γνωρίζετε ότι η αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρώπη έχει φτάσει σε ένα ε, πολύ σημαντικό επίπεδο ολοκλήρωσης. Αυτός ο χάρτης δείχνει τις δύο περιφερειακές αγορές που έχουμε. Έχουμε 18 κράτη-μέλη ε, και την Νορβηγία που πάμε από το ε, Γιβραλτάρ και από την θάλασσα, ως τη θάλασσα του Μπάρντ και μετά έχουμε την Τσεχία, Ρωμανία, Ουγγαρία και Σλοβενία. Επίσης έχουμε ζητήματα σχετικά με την Ιρλανδία και κάποιες άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν μπει ε, στη διαδικασία. Ε, ναι, δεν έχουν αγορά, αλλά υπάρχει σημαντική πρόοδος. Και αυτή η πρόοδος έχει ήδη δώσει καρπούς και ωφέλει στους καταναλωτές. Αυτό είναι το δικό μας, η δική μας εκτίμηση, αλλά ε, έχει να κάνει και γενικά με τους ε, διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς. Αυτό εκτιμούν και αυτοί. Έχουμε ένα ε, δις ετήσια ωφέλη. Έχουμε επίσης σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης, της δυναμικότητας διασυνοριακά. αν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ολοκλήρωση θα είχαμε άλλα 250 ε, εκατομμύρια το χρόνο ως όφελος. Τώρα, αν δούμε τι γίνεται την αγορά εξισορρόπησης που είναι και αυτή μια αγορά που θα μπορέσει να μας φέρει σημαντικά ωφέλη, γιατί μιλάμε για συμπληρωματική υπηρεσία για τις ώρες εχμής. Ε, αυτό μας φέρνει ε, ένα όφελος ετησίως γύρω στα 680 εκατομμύρια. Η αγορά των συμπληρωματικών υπηρεσιών, εάν ολοκληρωθεί πλήρως όλη την Ένωση, θα έχουμε άλλα τρία θα έχουμε τρία δις συνολικά όφελος. Τώρα, αυτά για τον ηλεκτρισμό. Για να δούμε τι γίνεται με το φυσικό αέριο. Αυτοί οι χάρτες δείχνουν τις διαφορές ε, στο sourcing cost σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή αυτό είναι το κόστος που πληρώνουν όταν θέλουν να αγοράσουν αέριο για να δώσουν στους πελάτες τους φαίνεται ότι αυτό το κόστος είναι ε, πολύ κοντά στο benchmark που έχουμε ε, για το TTF στην Ιρλανδία. Στο μπλε, στο βαθύ μπλε, έχουμε ακόμα μεγαλύτερες ε, διαφορές. 1 με 3 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το λευκό κομμάτι είναι αυτό στο οποίο έχει υπάρξει επέκταση και δεν είναι από τα ανατολικά προς τα δυτικά, αλλά πέρα από αυτό και γύρω από τη βασική αγορά που είναι στην Ολλανδία. Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός και η ολοκλήρωση είναι πιο σημαντική από την εγκύτητα στις πηγές. Η ευρωπαϊκή πολιτική λοιπόν για την ολοκλήρωση των αγορών ρευστότητας κυρίως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση κατά την άποψή μας λοιπόν. Υπό αυτό το πρίσμα ας αναφερθώ τώρα στις δραστηριότητές μας. Αυτές είναι στατιστικές. Είναι πολύ δύσκολο να χαρακτηρίσουμε τις δραστηριότητές μας με αριθμούς, αλλά να σας πω λίγο τι έχουμε κάνει σε επίπεδο γνωμοδοτήσεων, συστάσεων και αποφάσεων από το 2011. Ως τώρα και μέχρι πέρυσι ε, είχα, έχουμε καταθέσει 120 γνωμοδοτήσεις, 180 συνολικά, 120 είναι οι γνωμοδοτήσεις. Εμείς δεν έχουμε εξουσιοδότηση για να λαμβάνουμε αποφάσεις παρά μόνο για την εφαρμογή του REMIT θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Και πρόσφατα για τους όρους ε, και τις προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που έρχονται όχι μόνο για μας αλλά και για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Δεν θέλω τώρα να περάσω και να εξετάσω όλα τα σημεία αυτής της διαφάνειας. Αυτή η διαφάνεια συνοψίζει αυτά που έχουμε κάνει τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια. Απλώς για τα όσα θα ακολουθήσουν αξίζει να σας ε, μιλήσω λίγο για την δραστηριότητα παρακολούθησης της αγοράς. Από το 2012 εκδίδουμε κάθε χρόνο μία έκθεση η οποία εξετάζει την εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και τονίζουμε τις ζητήματα που προκύπτουν ή φραγμούς ε, στην αγορά. Είμαι σίγουρος ότι ήδη θα έχετε ακούσει ότι ένα από αυτά τα βασικά προβλήματα που έχουμε τώρα είναι ότι η ανταλλαγή διασυνοριακά ή μάλλον ε, η δυναμικότητα που διατίθεται για διασυνοριακές ανταλλαγές ε, ενέργειας ε, δεν είναι επαρκής έτσι ώστε να έχουμε μια ασφάλεια. Έχουμε αυτή τη λεγόμενη benchmark capacity. Τι είναι αυτό. είναι ας πούμε το συγκρίσιμο κριτήριό μας και εδώ βλέπετε ακριβώς πόσο είναι διαθέσιμο. Είναι περίπου το 50%. Άρα θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερες ε, διαθεσιμότητες. Σε κάποια σύνορα ε, είναι μικρότερο αυτό, 0-1-2% ε, ή ας πούμε Πολωνία προς Γερμανία, Τσεχία, σε άλλες χώρες 10% ή κάτω από το 10%. Ένας λόγος είναι ο τρόπος που, υπολογίζουμε τη δυναμικότητα. Είναι ας πούμε μια προσέγγιση τύπου λέγκαση. Ε, δηλαδή, αυτό που νοείται ως ε, δυναμικότητα είναι αυτά που εναπομένουν από τις ε, εξισώσεις για την ασφάλεια του συστήματος. Και όσον αφορά το επίπεδο συνεργασίας ε, μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Ε, εδώ έχουμε μια αδρή εικόνα, η οποία όμως λέει πολλά. Όπως βλέπετε, βάσει των απαιτήσεων του τρίτου πακέτου, ε, σε πολλές περιπτώσεις είμαστε κάτω από το 30% και συγκεκριμένα σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε κάτω και από το 10%. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε πολλά περισσότερα για να μπορέσει η αγορά να έχει τη δυναμικότητα για διασυνοριακό εμπόριο. Αν δούμε τώρα την αγορά αερίου, φυσικού αερίου, υπάρχουν και εκεί κάποιες προκλήσεις, γιατί έχουμε πολύ καλά ενεπτυγμένες αγορές, όπως ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ε, κάτω χώρες. Ήδη μίλησα για το TTF. Εκεί υπάρχει αρκετή ρευστότητα για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι ενδιαφερόμενοι, όμως ε, ε, σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει τέτοια πρόοδος. Η Σλοβακία και η Τσεχία, για παράδειγμα, περνάνε από το ένα επίπεδο στο άλλο, αλλά ε, πολλά έχουν να γίνουν ακόμα. Τώρα, όσον αφορά στο REMIT, που είναι Ε, ο κανονισμός ε, για την ολοκλήρωση και την διαφάνεια της αγοράς το 2011 ολοκληρώθηκε και δόθηκε η εντολή να υπάρχει μια ρυθμιστική εποπτεία των συναλλαγών, των εμπορικών συναλλαγών στον τομέα αυτό. Αυτό είναι ο τρόπος που το προσεγγίζουμε. Συλλέγουμε τα δεδομένα από το 2016, λαμβάνουμε εκθέσεις είτε για την ε, φυσική παράδοση είτε για τις οικονομικές, ε, οικονομικές συναλλαγές και διακανονισμούς. Μετά χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα alerts, δηλαδή συναγερμούς για κατάχρηση της αγοράς. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε κάτι τέτοιο μέσω αυτής της πληροφόρησης, όμως ε, κάποιες φορές μπορεί να είναι παράξενες οι συναλλαγές, αλλά να μην ενέχουν κατάχρηση της αγοράς. Αν λοιπόν αυτά μπουν στο αυτόματο σύστημα ε, αξιολόγησης ε, και διάγνωσης, μπορεί να έχουμε κάποια ανώμαλα συμβάντα, όπως ονομάζονται, αλλά αυτά ε, μπορούμε απλώς να τα περάσουμε στις ελληνικές ρυθμιστικές αρχές μόνο όταν θεωρούμε ότι υπήρξε παραβίαση του REMIT. Τώρα, το 2011 ε, ε, ξεκίνησαν αυτοί, αυτές οι απαγορεύσεις, από τότε έχουμε λοιπόν στοιχεία και να πώς ε, διαμορφώθηκαν οι υποθέσεις. Πέρυσι είχαμε 85 υποθέσεις ε, στις οποίες υπήρχε ενδεχόμενη παράβαση ως προς τον Ρέμιτ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα βέβαια σε επίπεδο πόρων και γι' αυτό έχουμε αυξημένο φορτό εργασία, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με όλε τι υποθέσει. έχουμε συσσωρεύσει πάρα πολλέ υποθέσει που δεν έχουμε εξετάσει. Έχουμε πολύ περισσότερο τέτοιο φόρτο από ό,τι είχαμε σε άλλα έτη. Αυτό είναι βέβαια φυσιολογικό, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτά τα επίπεδα. Για να δούμε τώρα τι ψάξαμε και τι βρήκαμε. Περισσότερες από τις πιθανές παραβιάσεις έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση της αγοράς και εσωτερική πληροφόρηση. Δηλαδή είναι διάφορες μορφές εκμετάλλευσης της αγοράς. Τώρα για τις προκλήσεις. Ίσως υπήρχε η αντίληψη κάποτε ότι σε επίπεδο σχεδιασμού της αγοράς ότι μόλις θα υιοθετούσαμε τον κώδικα και τα δίκτυα θα είχε γίνει περισσότερη δουλειά. Αυτό φαίνεται τελικά ότι δεν είναι αλήθεια γιατί ε, ο κώδικας αυτός ε, τελικά έγινε οδηγίες, κατευθυντήρες γραμμές ε, και υπάρχουν και άλλοι κανόνες πιο τεχνικοί που πρέπει ακόμα να αποφασιστούν. Είναι οι μεθοδολογίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις. Αν δείτε λοιπόν ακριβώς το forward capacity, το ignition balancing και το System Operation Balancing και έχουμε περίπου 200 τέτοιους όρους, προϋποθέσεις και μεθοδολογίες που ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί πέρα από τον κώδικα. Και αν δεν συμφωνήσουν οι εθνικές αρχές για αυτά, θα ε, έρθουν σε εμά οι υποθέσεις. Ως τώρα κάποιες ε, ε, υποθέσεις έχουν παραπευθεί σε εμάς και έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίληψη πλέον ότι το, ο κωδικός, η κωδική δικτύου θα μας κάνουν τη δουλειά. Για το φυσικό αέριο δεν έχουμε το ίδιο ε, καθεστώς, όμως πρέπει να κάνουμε εκθέσεις σχετικά με την, με, τα, με την εφαρμογή των κωδικών δικτύων. Έχουμε στοιχεία, θα τα ε, δημοσιεύσουμε και με χαρά μου θα επανέλθω για να σας μιλήσω για τα σημεία διασύνθεσης στο σύστημα αερίου Και ο τελευταίος ε, κωδικός ε, δικτύου ήταν για τις ε, τιμές. Θα θυμάστε τι ήταν αυτό. Ε, κυρίως είχε να κάνει με την διαφάνεια. Να μπορούν δηλαδή οι δημός οι εθνικοί ρυθμιστικές αρχές να δημοσιεύουν τιμές έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε και εκθέσεις σχετικά με το κατά πόσο οι μεθοδολογίες αναρμονίζονται με τα κριτήρια που έχουμε στον κώδικα. Εδώ είναι το προφίλ του εγγράφου διαβούλευσης που θα πρέπει να εξετάσουν φέτος οι αρχές. Βλέπετε ότι όλο το καλοκαίρι θα έχουμε πολλή δουλειά. 19 είναι το μεγαλύτερο νούμερο. 19 κωδικοί να εξετάζονται ταυτόχρονα και εγώ έχω μόνο τρία άτομα στην ομάδα για το φυσικό αέριο να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Τέλος για το REMIT, όπως ανέφερα, είναι μια διαδικασία με δύο στάδια. Πρώτον έχουμε αυτόματη ε, αυτόματη διαλογή. Έχουμε 45 με 50 χιλιάδες αρχεία συναλλαγών το μήνα που λαμβάνουμε και έχουμε 3.000 με 3.500 ε, ε, ανώμαλα περιστατικά το μήνα. Επειδή όμως ε, μπορούμε μόνο μέχρι 1.000 το πολύ να εξετάσουμε χειροκίνητα, καταλαβαίνετε ότι μόνο το 1 τρίτο μπορούμε να εξετάσουμε και στέλνουμε στις εθνικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές μόνο γύρω στα 50 το μήνα. Άρα χρειαζόμαστε περίπου 20 alert για να καλύψουμε όλους τους κοινούς τύπους κατάχρησης της αγοράς. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε μόνο 6 και μπορούμε να εξετάσουμε μόνο το 1 τρίτο της αγοράς. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να δώσουμε μια αξιοπιστή εικόνα, γιατί εξετάζουμε μόνο το 10% όσων έπρεπε να εξετάσουμε. Δεν λέμε βέβαια τι εξετάζουμε, έτσι ώστε αυτοί που συμμετέχουν στην αγορά να μην ξέρουν προς τα πού εξετάζουμε, σε ποια κατεύθυνση, αλλά από ό,τι φαίνεται πολλά απομένουν έτσι. Και τέλος, η τελευταία μου διαφάνεια, πριν ζητήσω από τον Γκάρετ να ολοκληρώσει στο πακέτο της ε, καθαρής ενέργειας δεν έχουμε προσωπικό σε δραματικά επίπεδα. Φέτος δεν είχαμε χρήματα για άδεια για το software και παρατρίχα να κλείσουμε και ένα σταθμό. Τελικά βρήκαμε αυτό το 1,5 εκατομμύριο που έπρεπε να βρούμε για του χρόνου. Αυτό που προτείνουμε είναι 31 ε, μία επιπλέον θέσεις, ε, ε, κυρίως για το REMIT. Αργότερα θα σας πω για το benchmark που δίνουμε σε σχέση με άλλα θεσμικά όργανα και άλλα 8 εκατομμύρια σε σχέση με αυτό που προτείνει η Κομισιόν για του χρόνου. Τα 4 εκατομμύρια θα είναι για το προσωπικό και τα υπόλοιπα θα είναι για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα χρήματα να πληρώσουμε για τις άδειες, ε, για το software ε, της ε, εποπτείας. Και εδώ δίνω το λόγο στον Γκάρετ για το τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ. Ναι, μια ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση. Δεν είναι εύκολο να την παρακολουθήσει κανείς βέβαια γιατί είναι πυκνή. έχετε το λόγο. Ελπίζω η δικιά μου να είναι πιο απλή να την παρακολουθήσετε η παρουσίαση γιατί θα μιλήσω για το μέλλον. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε έναν τόσο εργατικό και παραγωγικό ε, συντονιστή όπως ο Αλμπέρτο. Πρέπει να προχωρήσουμε όμως στο μέλλον οργανισμός μας θα αναλάβει και άλλα καθήκοντα, τα βλέπετε στην οθόνη. Θα έλεγα συνοπτικά ότι θα χρειαστεί να αναλάβουμε και άλλα καθήκοντα ακριβώς επειδή θα ε, άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί δεν έχουν επαρκείς αρμοδιότητες εποπτείας, εθνικές ρυθμιστικές αρχές Και αυτό θα συμβεί μέσω του φορέα μας και μέσω του πακέτου για την καθαρή ενέργεια. Η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πακέτο αυτό ήταν ε, εξαιρετική. Μας βοήθησε πάρα πολύ να ε, πάμε προς τα μπρος ως, ε, ως υπηρεσία. Καλωσορίζουμε όλες τις προτινόμενες διατυπώσεις που είδαμε από το Κοινοβούλιο σε κάποιες περιπτώσεις προκρίθηκαν οι διατυπώσεις και οι επιλογές του Συμβουλίου και ίσως να προτιμούσαμε κάτι διαφορετικό, γι' αυτό θα προσπαθήσω να σας εκθέσω αυτές τις απόψεις. Ε, το, πρόγραμμα, το πακέτο για την καθαρή ενέργεια είναι πολύ φιλόδοξο. Ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τις επιπτώσεις του θα τις ε, έχουμε στην υπηρεσία και γενικά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπετε τις λεπτομέρειες σας στην οθόνη, αλλά θα σας δώσω μια γενικότερη εικόνα. Αυτό που επιδιώκουμε με το πακέτο για την καθαρή ενέργεια είναι να προσθέσουμε και άλλα επιτεύγματα σε αυτά που ήδη πέτυχε και ήταν ήδη πολύ σημαντικά για την Ευρώπη, το τρίτο πακέτο για την ενέργεια. Νομίζω σε ένα στοιχείο στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι δεν υπήρχε το ίδιο επίπεδο φιλοδοξία. Το, το Κοινοβούλιο ήταν πολύ πιο φιλόδοξο. Η υπηρεσία μας λειτουργεί εδώ και κάμποσα χρόνια. Γνωρίζουμε ε, ότι στους τομείς εκείνους όπου έχουμε αποφασιστικές αρμοδιότητες τα πράγματα είναι δύσκολα. Και ένα στοιχείο που δυσκολεύει τη λήψη των αποφάσεων είναι η ομοφωνία που χρειάζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ΡΕΙ. Αν μία διαφωνή μπορεί να μπλοκάρει την απόφαση. Και αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο για εμάς γιατί έχουμε εκπροσώπους από τις ρυθμιστικές αρχές από όλη την Ευρώπη. Και, και, και διαπιστώνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε γιατί μία-δύο ρυθμιστικές αρχές διαφωνούν. Και ήθιστε αυτά τα θέματα στα οποία υπάρχει η έλλειψη ομοφωνίας να είναι τα πιο σημαντικά. Είναι δύσκολο 27-28 κράτη-μέλη και οι ρυθμιστικές τους αρχές να συμφωνούν για όλα τα θέματα. Μας ανησυχούν λοιπόν κάποιες από τις προτάσεις που βλέπουμε από το Συμβούλιο και ε, καλωσορίζουμε και προτιμούμε πολύ περισσότερο τις αντίστοιχες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αφορά τώρα τις νέες αρμοδιότητες και τις αποφάσεις που θα λαμβάνει με βάση αυτές πλέον η υπηρεσία μας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχει τη δυνατότητα κάποια θέματα να τα ρυθμίζει η υπηρεσία χωρίς να ρυθμίζονται όλα αναλυτικά στην νομοθεσία. Βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτιμά και επιθυμεί αυτή την διακριτική ευχαίρεια να την έχει η υπηρεσία. Αυτό είναι πολύ ε, πιο ευέλικτο αλλά και πολύ ορθότερο από πλευράς ποιότητας της νομοθεσίας η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι τεράστια ε, αγορά. Έχουμε τεράστιες αλλαγές επίσης. Έχουμε την εγκατάλειψη της χρήσης των τεχνολογιών του άνθρακα. Ε, πώς μπορεί κανείς σήμερα να προβλέψει ποιες θα είναι οι συνθήκες που θα ισχύουν σε αυτή την αγορά σε 5-10 χρόνια και να χρειάζεται κάθε φορά να αλλάζει με τις ε, αργές διαδικασίες την ομοθεσία. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την προσέγγιση που προκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι θα μας δώσει ε, μια καλύτερη θέση και την καλύτερη δυνατότητα να αντιποκρινόμαστε στις αλλαγές στο μέλλον. Ε, θα πρέπει η νομοθεσία να μας πηγαίνει προς τα μπρος, όχι να ε, οπισθοχωρούμε. Ένα από τα ζητήματα που έχει δημιουργήσει μια κάποια διαμάχη ε, και είναι φυσιολογικό, είναι η διάκριση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Διευθυντή της Acer και των Εθνικών ε, Ρυθμιστικών Αρχών. Θα σας παρουσιάσω την δύο πλευρές. Στον πίνακα αυτό βλέπετε με βάση το τρίτο πακέτο και την ενέργεια ε, για ποια ζητήματα μπορεί να λάβει απόφαση ο Διευθυντής και για ποια πρέπει να λάβει ε, την σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ε, το... Είναι σημαντικό και το βλέπουμε αυτό στο νέο νομοθετικό κείμενο του πακέτου για την καθαρή ενέργεια ότι χρειάζεται να έχουμε έναν, μια ισχυροποιημένη θέση για το διευθυντή, να μπορεί να έχει την πρωτοβουλία να θέτει προτάσεις σε εμάς, ε, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε τελικά να καταλήγουμε σε συμφωνία. Με μια διαδικασία συνενετική τελικά. Στο προηγούμενο προσχέδιο φαινόταν να υπονομεύεται κάπως η θέση του Διευθυντή, να του αποδίδονται περισσότερα, περισσότερο καθήκοντα συντονιστή, γραμματέα παρά Διευθυντή. Πρέπει να γίνουν προσεκτικές επιλογές για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η σχέση. Και μιας και είναι και παρόν ο Διευθυντής, ίσως θα μπορούσε να το πει και ο ίδιος, Ωραία, καλύτερα να το συζητήσουμε μετά. Επίσης ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το, η συλλογή τελών για την υπηρεσία άμεσα από τις ε, επιχειρήσεις του κλάδου και μπορώ να σας μοιραστώ την εμπειρία μου που, όπου στην Ιρλανδία η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή έχει αυτό το δικαίωμα και είναι πολύ μεγάλη εξουσία και πολύ μεγάλο, έχει πολύ μεγάλη σημασία για το σεβασμό της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής να μπορεί να επιβάλλει τέτοια τέλη άμεσα στη βιομηχανία, χωρί να χρειάζεται να περάσει από τη γενικότερη διαδικασία του προπολογισμού που πρέπει να βρει ισορροπίε ανάμεσα και σε άλλε πολιτικέ προτεραιότητε που έχει η εκπαίδευση η υγεία. Και αυτό θα έχει μεγάλη σημασία και για την Ευρωπαϊκή Αντίστοιχη Υπηρεσία. Βεβαίω θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Ε, τα τέλη αυτά θα πρέπει να εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Διοικητικό Συμβούλιο, φυσικά. Όμως, ίσως θα είχε επίσης νόημα να δούμε εάν τα τέλη αυτά θα μπορούσαν να επιβάλλονται σε περισσότερα είδη φορέων. Κάτι τέτοιο θα δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες στην υπηρεσία μας. Κλείνοντας, τελευταία διαφάνεια, ήθελα να κάνω και λίγη διαφήμιση, γιατί στις 5 Ιουλίου διοργανώνουμε ένα συνέδριο και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, σας προσκαλώ ιδιαίτερα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να ακούσουμε τις δικέ σας απόψει όχι μόνο τι απόψει του κλάδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Βλέποντας εδώ το πολυάριθμο πλήθος, δύο από τους συναδέρφους έχουν ζητήσει το λόγο. Ο πρώτος, μια που μιλήσατε και για την Ιρλανδία, είναι ο συνάδελφος Σον Κέλλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Είναι όντως πολύ σημαντικό για μας με τις συζητήσεις που γίνονται αυτή την εποχή και σας άκουσα προσεκτικά. Αναφερθήκατε στους ελέγχους και στο θέμα των διαφόρων αξιωμάτων και του συναδέρφου που έχει ανέλθει. Μπορείτε να προχωρήσετε, γιατί πολλές φορές οι μικρές χώρες είναι που κάνουν τα θαύματα. Και εν ώψη του Brexit το ρυθμιστικό πλαίσιο που αναφέρεται για το πακέτο για την καθαρή ενέργεια. Εγώ ήμουνα από το ΕΛΚΑ εισηγητής και έχουμε κάνει διάφορους τριμερείς διαλόγους. Συνεχίζουμε και αύριο μετά τη συνάντηση με τους κοιόδες εισηγητές που είχαμε χτες. Και η ενισχυμένη φιλοδοξία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό από κάθε άποψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μεταξύ άλλων, πιέζοντας το Συμβούλιο να προχωρήσει. Γιατί υπάρχει απροθυμία στο Συμβούλιο να προχωρήσει γρήγορα. Εξού και η μεγάλη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μπορούμε να δούμε τα πράγματα κάπως πιο αντικειμενικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να φροντίσουμε για προτάσεις που να έχουν πραγματικά νόημα. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να καταλήξουμε και για το πακέτο αυτό για την καθαρή ενέργεια. Και εσείς έχετε να παίξετε σημαντικό ρόλο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα τα καταφέρουμε. Θα προχωρήσουμε μαζί και θα υπάρξουν και οι κατάλληλοι πόροι ώστε να υλοποιηθεί το πακέτο αυτό με τον τρόπο και έτσι όπως το προετοιμάσαμε και τον κρίναμε. Ίσως θα πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα ή εμείς να πιέσουμε ως ευρωβουλευτές το Συμβούλιο ακόμα περισσότερο. Να ξέρετε ότι έχετε ένα σύμμαχο εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητές συνάδελφε για τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Φέντερλε, εκ μέρους του κύριου Πέτερσον, που είναι ο εισηγητής για το ΑΣΕΡ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, ο κύριος Πέτερσον ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα, αλλά χρειάστηκε να επιστρέψει στην ε, Δανία. Εκ μέρους του όμως θέλω να ε, σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία, έτσι λέει ο κύριος Φέλλερ, ότι είχε πολύ καλή συνεργασία μαζί σας. Και θέλει να υπογραμμίσει την καλή δουλειά που, και την καλή συνεργασία που είχε με τον κύριο ήταν πάρα πολύ σημαντικό το έργο του Διευθυντή. Και υπογραμμίζει επίσης ότι η ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όντω χρειάζεται έναν οργανισμό που να μπορεί να ελέγχει, να εποπτεύει το τι γίνεται στην αγορά, ώστε να υπάρξει παρετέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η ολοκλήρωση αυτή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια και προκειμένου να έχουμε εναλλακτικέ μορφές ενέργειας παντού στην Ευρώπη. Επίσης εκφράζει την ικανοποίησή του με τον συμβιβασμό ο οποίο ε, πετεύχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΑΣΕΡ χρειάζεται και άλλα μέσα για να μπορέσει να τελέσει πλήρως και το σκοπό του. Περισσότερους πόρους, και δεδομένου ότι έρχεται από το βορρά, χαίρεται που δεν θα υπάρχουν διακρίσεις για την ενέργεια από άλλες χώρες μέλη. Και κύριος Κέλλη σωστά λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να τοποθετηθεί όσον αφορά την ενεργειακή αγορά ακριβώς γιατί έτσι καλώς εμείς έχουμε εθνικές τέτοιες εταιρείες, άρα δεν έχουμε ίδιο συμφέρον. Χαίρομαι πάντως που η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπέρ των καταναλωτών και του κλάδου στην Ευρώπη. Ακριβώς για το όπως λέτε και εσείς, εμείς βλέπουμε τα πράγματα από κάποια απόσταση, όχι όπως οι χώρες μέλη στο Συμβούλιο. Πρέπει η ενέργεια να κυκλοφορεί ελεύθερα όπως και άλλες υπηρεσίες και αγαθά. Στις προεκλογικές εκστρατείες ορισμένοι λένε ότι έχουμε υπερβολική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελάχιστες μοναδιές, ε, μοναδιές πόρους. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό. Μια ευρύτερη αγορά θα είχε όφελος για όλες τις χώρες. Ο προστατευτισμός έχει εμποδίσει την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, ακόμα και αν πέφτουν οι τιμές της ηλιακής και της ολικής ενέργειας ο κύριος Πέτρος ζητάει από τις χώρες μέλη και το Συμβούλιο να φροντίσουν να τηρηθούν οι υποχρώσεις που αναλάβαμε στο Παρίσι. Ξέρουμε ότι αυτό δεν προχωράει αρκετά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό που το ζητάει επίμονα λέει ο κύριος Πετσέλη ότι είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί εκ μέρους των Ευρωπαίων καταναλωτών και μας ζητάει να επιδείξουμε θάρρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Ναι, και εγώ είμαι πεπισμένος ότι θα συναντηθούμε με τον κύριο Ποτότσνικ ξανά πριν αλλάξει ιδιότητα στον ΑΣΕΡ. Ε, ευχαριστούμε για αυτά που είπατε κι εσείς. Ελπίζω το Σεπτέμβριο, το πολύ τον Οκτώβριο να ξανασυναντηθούμε. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Όλιβερ Κόχ που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει και εκείνο την άποψη της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΑΣΕΡ σίγουρα αξίζει την ίδια προσοχή όπως το Brexit που συζητήσαμε πριν. Δεν θα μπορούσε κανείς να υπογραμμίσει αρκετά πόσο ρόλο κλειδί παίζει η ΑΣΕΡ για την εσωτερική αγορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε μόνο τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή με το Brexit ε, ακούσαμε για αυτά τα προβλήματα που ανέφερε και ο Διευθυντής. Τέτοια πράγματα όμως προκύπτουν κάθε 2-3 χρόνια και κάθε 2-3 χρόνια ο κόσμος συνειδητοποιεί το ρόλο που παίζει ο Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστών Ενέργειας, ο ΑΣΕΡ. Τα Πατότσνικ και η ομάδα του που θα άξιζε ένα βραβείο πραγματικά για τα όσο καταφέρνει για την εσωτερική αγορά. Μας είπε λοιπόν ότι η εσωτερική αγορά φέρνει τεράστια ωφέλη και ασφάλεια εφοδιασμού που δεν θα είχαμε χωρίς να μπορούμε να έχουμε περισσότερα. Λοιπόν, οι καταναλωτές και η Ευρώπη ξοδεύουν πολύ περισσότερα χρήματα ακριβώς επειδή δεν έχουμε την ολοκλήρωση της αγοράς. Και τώρα με το Brexit πρέπει να αποφύγουμε επιπλέον ο κόστος εξαιτίας της μη λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Θα μπορούσε να συνεχίσει ο κύριος Ποτότσιν για μισή ώρα, για ώρες τέλος πάντων, να δείχνει τα εμπόδια που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά ακόμα και που μας εμποδίζουν να επωφεληθούμε πλήρως. Κάτι το οποίο κοστίζει χρήματα στη... στους πολίτες. Φραγμή στα σύνορα, για παράδειγμα. Ε, αυτά είναι πράγματα για τα οποία χρειαζόμαστε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τους επόμενους μήνες. Ο κύριος Ποτότσνικ παρουσίασε την κατάσταση που είπε το 50% των διασυνοριακών ροών κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά αλλού, μόνο στον ηλεκτρισμό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η διαδικασία δεν είναι εύκολη για να συμφωνήσουν οι χώρες μέλη για τον κανονισμό ΙΖΑ. Είναι ο μόνος κανονισμός όπου το Συμβούλιο δεν κατάφερε να υιοθετήσει ούτε καν μια γενική προσέγγιση. Ελπίζουμε αυτό να διορθωθεί σε λίγες μέρες. Πάντως, ο, το καθήκον του ΑΣΕΡ θα είναι πολύ σημαντικό και στο μέλλον. είναι πολύ βασικό να αναγνωρίσουμε ότι ο ΆΙΣΕΡ δεν είναι απλώς ένα όργανο, αλλά αποτελεί ένα βασικό στοιχείο, ένα συνδετικό κρίκο. Χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος συντονίζει, ελέγχει. Αν το χάσουμε αυτό, τότε θα έχουμε τεράστια εμπόδια. Και γι' αυτό από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ανησυχούσαμε πάρα πολύ αν δεν αναγνωριζόταν πλήρως ο ΑΣΕΡ και αν με το πακέτο του 2009 αντί να πάμε μπροστά πήγαμε πίσω. Είπατε ότι σε κάποιες προτάσεις υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που κυκλοφορούν που θα πήγαιναν το ρολόι πίσω. Ελπίζουμε στους τριμερείς διαλόγους, στο δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς αυτής, να βρούμε λύσεις που θα το εμποδίσει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προτάσεις με μικρή ενίσχυση του ρόλου του ΑΣΕΡ. Πολύ θα το θέλαμε. Πρέπει πάντως να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η συζήτηση για τον ΑΣΕΡ είναι στοιχείο κλειδί για τη λειτουργία της αγοράς. Ελπίζουμε να έχουμε τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε για τον βασικό ρόλο που παίζετε ο οργανισμός σας. Για μας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Και αυτό και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσίαση και προσβλέπουμε σε παρετέρω συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χοχ. Θέλετε να κάνετε και κάποια σχόλια τώρα για αυτές τις ε, ερωτήσεις. Α, ο κύριος Λάγκεν, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στην παρουσίαση, τη διάβασε και τώρα έχει κάποιο σχόλιο να κάνει. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ήρθα πολύ αργά, διότι δυστυχώς η εικόν και η ε, οι δύο επιτροπές μου λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. Άκουσα όμως ε, όλα όσα έχουν παρουσιάσει οι ομιλητές, ειδικά ο κύριος Κόχα, φαίνεται ότι έχετε κάνει μια πολύ καλή δουλειά και όσον αφορά στην κοινή θέση του Κοινοβουλίου για την αλλαγή του κανονισμού ΕΣΕΡ στις 26 Φεβρουαρίου έγινε αυτό, ε, τότε πήραμε αυτή την απόφαση και έκτοτε δεν ε, ακούσαμε τίποτα από το Συμβούλιο. Δεν ε, είχαμε ούτε μία κίνηση από την πλευρά του Συμβουλίου. Θα ήμουνα λοιπόν πραγματικά ε, ευγνώμων κύριε Αντιπρόεδρε αν λέγατε στον πρόεδρο Μπούζεκ ότι πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Δεν μπορούμε να μην έχουμε πρόοδο γιατί δεν το θέλει το Συμβούλιο και πραγματικά η Βουλγαρική Προεδρία μας ε, ε, έχει εξασθενήσει τη θέση μας. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το τριμερή διάλογο. Όπως είπε ο κύριος Κοχ, θέλουμε μια βελτίωση. Δεν θέλουμε όλα όσα θέλουν στο ΆΣΕΡ. Είμαστε κάτω και από τις προσδοκίες της Κομισιόν, αλλά θέλουμε μια καλύτερη ας πούμε, δυναμική και πραγματικά ε, στο Κοινοβούλιο ε, δεν θέλουμε πραγματικά λίγο πριν τις επόμενες ευρωεκλογέ ε, να διαπιστώσουμε ότι δεν θα υπάρχει σωστή ομοφωνία εδώ. δεν το αξίζει ο Άσερ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. λαμβάνω υπόψη τα σχολεία σας. Θα τα διαβιβάσω στον κύριο Μπούζεκ φυσικά και αύριο θα τον δείτε και προσωπικά. Θα διατρανώσουμε αυτή την άποψη και να δούμε τι να κάνουμε. Να πάμε λίγο ε, και την ε, οδηγία για το αέριο πιο μπροστά. Είναι ένα χρόνο η καθυστέρηση. Ωραία. Κύριε Ποτέσνικα, έχετε τώρα το λόγο και εσείς και ο κύριος Μπέρνου για να κάνετε σχόλια σχετικά με τόσα είπαν οι ευρωβουλευτές. Να σας ευχαριστήσω όλους ε, για την υποστήριξη στον οργανισμό. Να μιλήσω λίγο στο φίλο μου τον Ιρλανδό στην γλώσσα μας. <laughs> Θα περιορίσω τη χρήση της Ιρλανδικής σε αυτό. Ο κύριος Ποτόσνικ βέβαια δεν θα ξαναπεί διάφορα, ε, δεν θα κάνει μια παρουσίαση, θα πει απλώς ε, πόσο πραγματικά Χαιρόμαστε που έχει δημιουργηθεί ο οργανισμός, που έχει αυτή την ε, επιτυχία και είμαστε ευγνώμονες για όλα αυτά. Ναι, να πω κι εγώ κάποια σχόλια. Ευχαριστώ καταρχάς τον κύριο Κέλλη, τον κύριο Λάγκεν και τον κύριο Φέτερλη για τα ευγενικά τους λόγια για τον οργανισμό μας. Το Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή έχουν υποστηρίξει το έργο μας και σε δημοσιονομικό επίπεδο αλλά και τη δουλειά που κάναμε δόθηκε προσοχή μεγάλη. Ο κύριος Πέτερσιν ήρθε δύο φορές στη Λουμπλιάνα και πραγματικά και στις δύο συναντήσεις είχαμε πολύ επικοδομητική συνεργασία και πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τα όσα έχουμε κάνει για το πακέτο για την καθαρή ενέργεια αυτό ε, ξεπληρώνει κάπως τη δουλειά που έχουμε κάνει. Δεν υπήρχαν ερωτήσεις, οπότε τα τρία λεπτά που μας μένουν θα μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω για δύο σχόλια. Καταρχάς ο Γκάρετ αναφέρθηκε σε κάτι που έχει να κάνει ε, με τη δυναμική μεταξύ, στη σχέση μεταξύ του Συμβουλίου και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Το Συμβούλιο προσπαθεί να αλλάξει αυτή τη δυναμική. Μία από τις διαφάνειες που παρουσίασε ε, ο Γκάρετ είναι ακριβώς αυτή η σχέση του Συμβουλίου των Ρυθμιστικών Αρχών που δίνει κάποιες γνωμοδοτήσεις. Ε, όμως κάποια πράγματα δεν απαιτούν τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Βέβαια, εμείς ε, συζητάμε τα πάντα. Η διαδικασία συμπεριλαμβάνει τα πάντα, αλλά τελικά κάποιες ε, από τις δραστηριότητες του οργανισμού γίνονται με τον τελικό λόγο του ε, διευθυντή. Και ένα από τα βασικά στοιχεία που συμβαίνει αυτό είναι η έκθεση παρακολούθησης της αγοράς ε, που την παρουσιάζουμε κάθε χρόνο και εξετάζει τι συμβαίνει στα διάφορα κράτη-μέλη. Βρίσκει τα προβλήματα, τους φραγμούς, τις καθυστερήσεις, την μη συμμόρφωση. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία του οργανισμού έναντι των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για να μπορεί αυτή η έκθεση να δίνει μια αξιόπιστη και πραγματική εικόνα για τα όσα συμβαίνουν. Προσπαθώ πάντοτε να ακούω όλα τα μέλη του Συμβουλίου του Ρυθμιστικού Συμβουλίου τέλο πάντων, αλλά ε, η εικόνα που τελικά πρέπει να δώσουμε πρέπει να είναι η πραγματικότητα και θα είναι τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα εάν αυτό το Συμβούλιο έπρεπε να ευχαριστήσει τους πάντες, δηλαδή τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Ε, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα που δεν τους αρέσει να ακούνε, αλλά και προς δικό τους όφελος τελικά. Η διαμόρφωση του υφεστάμενου κανονισμού, δηλαδή ε, ο τρόπος που ρυθμίζεται η σχέση μεταξύ ε, του Διευθυντή και του Συμβουλίου είναι σωστή. Έχουμε το ρόλο εκείνου που καταδεικνύει τα προβλήματα και τις βέλτιστες πρακτικές. Γιατί το ο οργανισμός μας ε, πρέπει να διασφαλίσει την ε, εφαρμογή με συνεπή τρόπο και συνεκτικό τρόπο του κανονισμού. Τώρα, να αναφερθώ και σε κάποια άλλα ζητήματα που μας έχουν ανατεθεί. Ανέφερα για πολλές φορές το benchmark που έχουμε με την FEDRC, την ε, Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ρύθμισης ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, χρησιμοποιούν τρεις φορές περισσότερους πόρους για αυτούς από ότι θα, έπρεπαν, θα έπρεπε. Γι' αυτό δεν είναι δίκαιο ούτε για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Θα πρέπει οι τιμές να μην στρεβλώνονται από κατάχρηση και χειρισμό της αγοράς. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία εμείς κοιτάμε. Αν μου λέγανε να σταματήσω με το Remit, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα γιατί θα κοιμόμουν περισσότερες ώρες ε, τη νύχτα, αλλά το οφείλω στους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, υποστήριξη. Ίσως αυτή να είναι και η τελευταία φορά που με βλέπετε, δεν ξέρω. Ευχαριστώ και την Κομισιόν γιατί ήταν εταίρος μας ε, σε αυτόν τον δρόμο γεμάτο εμπόδια. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τα όρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη, ειδικά ως προς τη διαθήκη βορρα βορρά-νότου, του αγωγούς φυσικού αερίου και φυσικά τις γραμμές, τις συνδετήριες γραμμές που δεν χρησιμοποιούνται. Δεν είναι νέες πληροφορίες, γνωρίζουμε τα προβλήματα και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ξεκάθαρα, τα έχουμε στο μυαλό μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την αναφορά σας, στη συζήτηση. Σας υποστηρίζουμε συνεχώς ε, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο προς την ε, κατανομή των πόρων δικαίως ε, για τους ανθρώπινους πόρους και μη ανθρώπινους πόρους. Όσον αφορά στο τριμερή διάλογο, η Ήτρε έχει μια εντολή για να διαπραγματευτεί που θα διασφαλίσει έναν ισχυρό ρυθμιστικό ρόλο για τον οργανισμό σας. Μετά από αυτό να σας ανακοινώσω αγαξιότιμοι συνάδελφοι ότι έχει ακυρωθεί η συνεδρίαση για αύριο το πρωί. Θα ξεκινήσουμε στις 3 ε, το μεσημέρι αύριο μέχρι τις 6.30 το απόγευμα για την επιστήμη και την καινοτομία ε, και το πόσο ανοιχτές είναι στον κόσμο. Μιλάμε για ένα ε, πρόγραμμα συνεργασίας με το ΣΤΟΑ και το STS Forum. Να θυμάστε λοιπόν ότι το πρωί είστε ελεύθεροι να πάτε και να συμμετάσχετε σε όποια δραστηριότητα θέλετε. Το απόγευμα από τις 3 θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.